Good afternoon everyone. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρώτα πρώτα έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Φαντάζομαι ότι εγκρίνεται. Δύο έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 7ης Μαΐου και της 8ης Μαΐου. Από ό,τι βλέπω, ξέρω δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με αυτά. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Τρία. Is, ε, announcement, first announcement. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτον, η αλλαγή της αίθουσας για αύριο. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσουμε στο 5G3. 5G3. Αυτό λόγω του φόρτου εργασίας. Δεύτερη ανακοίνωση. Προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για την έλλειψη προόδου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή δημοσιονομικές υπηρεσίες. Οι συντονιστές αποφάσισαν την περασμένη Πέμπτη στο, στο Εστρασβούργο να κατατεθεί προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο για την έλλειψη προόδου για τις δημοσιονομικές και χρηματοστατικές υπηρεσίες και άλλες καθυστερήσεις. Τα ερωτήματα αυτά θα συνοδεύονται και από δύο-τρία ψηφίσματα, από ένα-δύο ψηφίσματα στον Ολομέλεια του Ιουνίου οι προφορικές ερωτήσει προς το Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον τρει εβδομάδες πριν την Ολομέλεια που πρέπει να απαντηθούν. Και επειδή επήγε το θέμα, οι συντονιστέ συμφώνησαν το προφορικό ερώτημα στο Συμβούλιο να κατατεθεί αμέσως. Και γι' αυτό ο πρόεδρος Μπόουλ την κατέθεσε εξ ονόματος της Οικονομικής Επιτροπής. Θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη και το ψήφισμα ετοιμάζεται. Τελευταία ανακοίνωση. Ο τριμερής διάλογος για το στατιστικό πλαίσιο, για την κανονισμό του στατιστικού πλαισίου. Στην πρώτη συνεδρίαση το θέμα συζητήθηκε στο σύνολό του και καθώς και οι διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες βρίσκουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται και αυτά που, δημοσιεύει το Eurostat. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 3 Ιουνίου. Τώρα λοιπόν περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την εξέταση των τροπολογιών για την έκθεση υποδηματά Θέσπιση ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δίνω λοιπόν αμέσω το λόγο στην κυρία Υποδηματά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και για τη δουλειά τους. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω την νομοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η Επιτροπή και ο συγγετής ο κ. Παλμιέρη έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και υποστήριξαν τη θέση μας για το φορό χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στη συζήτηση των τροπολογιών της εκθεσής μου. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι κατόπιν τριών ετών έντονων προσπαθειών με ηγετικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε τώρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία από 11 κράτη-μέλη για την εισαγωγή του φορού χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το Κοινοβούλιο είχε αυτό το θέμα σε υψηλή προτεραιότητα και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για να πείσει την Κομισιόν να τροποποιήσει τη θέση της και να προωθήσει μια νομοθετική πρόταση. Αυτό έγινε λοιπόν. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο όλοι έχουμε δει ότι υπήρξε μία έντονη εκστρατεία λόμπινγκ για να αποδυναμωθεί η πρόταση, μάλιστα και για να καταργηθεί εντελώς. Ε, νομίζω ότι αυτές είναι δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας στρατηγικής. Εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, καθώς ε, εισάγουν πάρα πολλές εξαιρέσεις, δημιουργούν νομικά κενά και επιτρέπουν ε, κάποιες προνομιούχες ε, λύσεις. Έτσι λοιπόν δε, αυτό δεν θα επέτρεπε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο φόρος και θα οδηγούσε σε αποτυχία του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όπως μας έχει δείξει η εμπειρία της εθνικής εφαρμογής του φόρου αυτού συγκεκριμένα στη Σουηδία. Επομένως, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αργό θάνατο του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αντί για έναν αφινιδιό θάνατο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο κατέβαλε προσπάθειες για την εισαγωγή αυτού του φόρου, δεν μπορεί τώρα να ειδωθεί ότι προωθεί εξαιρέσεις για το φόρο, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε καθόλου να συνάδει με το προηγούμενο έργο μας. Τώρα είναι η στιγμή να υποστηρίξουμε το φόρο και να αντισταθούμε σε απόπειρες του. Να έρθουμε τώρα στις τροπολογίες. Έχουμε λάβει 150 τροπολογίες, οι περισσότερες κατατέθηκαν από λίγους συναδέλφους και κυρίως από μη συμμετέχουσες χώρες που ζητούν εξαιρέσεις. Υπάρχουν και τροπολογίες που ε, ζητούν νόμιμα, νόμιμες ενσυχίες. Ε, να εισαχθεί αυτό το θέμα. Εμεί δεν θέλουμε να υποσκάψουμε το να καλύπτει ο φόρος όλες τις χρηματαγορές, όλα τα προϊόντα και όλους τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Οι τροπολογίε 96, 102, 104, 106, 114 καλούνται εξαίρεση των συνταξιδοτικών ταμείων λέγοντας ότι ο φόρος θα έχει επίπτωση στα έσοδα των συνταξιούχων. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ποινικοποιηθούν οι συνταξιούχοι, το αντίθετο. Τα συνταξιδοτικά ταμεία θα προσαρμόσουν τις εργασίες τους και θα στραφούν προς κάποιες πιο συντηρητικές στρατηγικές και αυτό θα ωφελήσει τους ίδιους τους συνταξιούχους και την οικονομία συνολικά. Το καθήκον των συνταξιοδοτικών ταμείων είναι να επενδύουν σε αποταμιεύσεις και να τις επιστρέφουν μετά από 20-30 χρόνια. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στο λεπτό θέμα ε, της φορολόγησης που τίθεται στις τροπολογίες 95 116-117 μπορεί ε, να υπάρχει κάποια παρεξήγηση σε σχέση με τη φορολόγηση πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς κρατικών ομολόγων. Αυτή είναι η κύρια αγορά που καθορίζει το κόστος ε, των κρατικών ομολόγων και είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή. Έτσι λοιπόν ένας επενδυτής με μία καθολική στρατηγική θα αγόραζε στην πρωτογενή αγορά όπου δεν υπάρχει φόρο και καθώ αναμένεται οι περισσότεροι επενδυτέ να στραφούν στις πρωτογενείς αγορέ, ο ανταγωνισμό, πιστεύω θα σκίσει μία πίση προ τα κάτω στο κόστο τη χρηματοδότηση. Αν υπήρχε στι πρωτογενεί αγορές ε, λόγω του χρεοφόρου χρηματιστικών συναλλαγών στι δεύτερογενεί αγορέ, ε, αυτό θα αντισταθμιζόταν από τα έσοδα από το φόρο, σύμφωνα με εκτιμήσει ε, τη Κομισιόν. Υπάρχει όμω ένα ζήτημα. Αν τα έσοδα έξοδα από αυτά τα ομόλογα θα καταναμηθούν ε, όπως πρέπει, δικαίως δηλαδή, μεταξύ των 11 κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να επιληθεί αν λόγου χάρη εφαρμόσουμε την αρχή της έκδοσης ε, καταρχήν και όχι στο τέλος ε, στην περίπτωση αυτών των κρατικών ομολόγων και Κάτι τελευταίο, μία εξαίρεση του κρατικό ομολογό θα δημιουργούσε άδικη μεταχείριση έναντι άλλων προϊόντων όπως τα εταιρικά ομολογά. Όμως καταλαβαίνοντας την ε, ευαισθησία του θέματος προτείναμε και άλλη λύση στους σκιώδεις εισηγητές να μπει μία αναφορά στη αναθεώρηση για να είμαστε σίγουροι ότι ο φόρος για ε, τα κρατικά ομολόγα θα μελετηθεί εκ του σύνεγγυς και επίση είμαι ανοιχτή να συζητήσω και να εισαγωγώ μία προσωρινή ρήτρα διασφάλισης στην περίπτωση το spread ενός τέτοιου ομολόγου φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δέκα τροπολογίες περίπου καλούν εξαίρεση των market makers στο πεδίο εφαρμογή των ε, αξιώσεων του φόρου. Γιατί εγώ να σας πω ότι οι market makers ε, ουσιαστικά εμπορεύονται για το δικό τους λογαριασμό και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τους εξαιρέσουμε από το φόρο πιστοτικών συναλλαγών καθώς δεν ε, επιτελούν δημόσια υπηρεσία αλλά κερδίζουν από την εμπορία. Αν εξαιρεθούν τότε κάποιοι τέτοιοι θεσμοί που έχουν εγγραφεί ως market makers Οπότε θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την εμπορία χωρίς να φορολογούνται. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα δημιουργούσε ένα νομικό κενό που θα διαστρέβλωνε την αγορά. Δεύτερο, αν τους εξαιρέσουμε, θα προσφέρουμε εξαίρεση και σε εμπορία υψηλή συχνότητα. Επίσης υπάρχει η διαχείριση των ρευστών, στη οποία, το θέμα το οποίο θίγουν έξι τροπολογίες και αυτό σχετίζεται με τις συναλλαγές εντός του ομίλου σε δέκα τροπολογίες αναφέρεται αυτό και από ό,τι καταλάβει η κυρία ανησυχία είναι το πρόσθετο άχθος ε, για το σεβασμό των απαιτήσεων που έχουν σεχθεί από την Οδηγία Κεφαλικών Οικοτήσεων 4 και της DRR. Επίσης πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις της αγορές ρέπο. Η διαχείριση των αγορών ρευστών είναι κάτι ευπρόσδεκτο και εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν εγγυημένα δάνεια, όμως προκειμένου να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες θα πρότεινα ένα χαμηλότερο ποσοστό για τα βραχυπρόθεσμα ρέπος μέχρι τους τρεις μήνες στο επίπεδο του 0,01% αντί για 0,1%. Αυτό θα καθιστούσε την αγορά οικονομικά βιώσιμη. Να τονίσω ότι αυτό θα είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς το 17% είναι ε, αγορών που φτάνουν τα 3, ε, 6 ε, Είναι κάποιες συναλλαγές πολύ συχνές και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ευνοούσε και τα συντοξιδοτικά ταμεία, που έχουν αποθεματικά και παραδοσιακά ε, προβαίνουν σε συναλλαγές ρέπο, έτσι ώστε θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα χωρίς υπερβολικό κίνδυνο. Να αναφερθώ σε κάποιες άλλες τροπολογίες που έχουν ε, να κάνουν με τις νόμιμες ανησυχίε. Έχουμε την τροπολογία 38 που καλεί τα κράτη-μέλη να ε, αναθεωρήσει οποιαδήποτε τραπεζική νομοθεσία έχει εισαγάγει τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ε, ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στην ε, τροπολογία 97 έχουμε το θέμα των μη χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων και καθώς αυτός ο φόρος απευθύνεται στο χρηματοπιστωτικό τομέα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν παράπλευρες απολύσεις για να μειώσουμε αυτές τις συνέπειες στην πραγματική οικονομία προτείνουμε να καλύπτουμε ε, κοιήτες μη χρηματοπιστικές συναλλαγές αν είναι κερδοσκοπικές. Ε, και στην τροπολογία 52 των κυρίο Κάρας Παλώνεν και Πιετικά είναι, την υποστηρίζω, εκεί ζητούνται μεγαλύτεροι συντελεστές της εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο Ζαν Πολ Γκοζές και ο Ζαν Πολ Μπεσέτ με την τροπολογία 74 και την τροπολογία 79 αναφέρονται στις currency spot transaction. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εισαχθούν εντό του πεδίου εφαρμογή κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο κύριος Κλούτα έχει εισαγάγει τις τροπολογίες 94 για την 149, για την ε, μεγάλη κερδοσκοπία ε, στις αγορές εμπορευμάτων, αγαθών. Και, αυτή είναι καλή, και αυτές οι τροπολογίες είναι καλές. Και να πω κάτι για το θέμα των ιδίων πόρων πριν κλείσω ο Μαρκάρα και Ζων Μπεσέτ στις τροπολογίες 29 και 31 έχουν εισαγάγει την ιδέα να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα του φόρου ως πρόσθετη είδη πόρη χωρίς ε, μείωση στην ε, συνεισφορά που γίνεται βάση του ακαθαρίστου εγχώριου εισοδήματος. Εγώ αυτή την ιδέα τη θεωρώ επί της αρχής θετική, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θα ήταν δίκαιη υπό την διαδικασία αυτή που ακολουθείτε τη ενισχυμένη συνεργασία για τα 11 κράτη-μέλη, γιατί θα συνεισφέραν ε, αναλογικά πιο υψηλά σε ένα προπολογισμό που έχει σχεδιαστεί για 27 κράτη-μέλη. Για τους λόγους αυτούς η πρότασή μου είναι να υποστηρίξουμε την ιδέα των πρόσθετων ίδιων πόρων όταν και τα 27 κρατημέλη θα συμμετέχουν στο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και το τελευταίο συμπερασματικό σχόλιο να υπενθυμίσω ότι η ευρεία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο συμφώνησε ότι ο χρηματιστοτικό τομέα είναι ένα τομέα που υποφορολογείται και ότι ο φόρο χρηματιστικών συναλλαγών είναι το σωστό εργαλείο για να διορθωθεί αυτή η ανισορροπία. Α δούμε προσεκτικά τι πιθανέ αρνητικέ συνέπειε. Όμω, να σεβαστούμε ταυτόχρονα τον, ε, το ευρύ πεδίο εφαρμογή για να πετύχει ο φόρο. Και όπω ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι συνομοθέτης ε, για την πρόταση αυτή. Αλλά η θέση μας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτικά. Αν πούμε όχι σε αυτή την ερχιστρωμένη προσπάθεια να προωθηθούν διάφορα είδη εξαιρέσεων, πιστεύω ότι θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο, ότι περιμένουμε από αυτού να τηρήσουν τι δεσμεύσει και τι υποσχέσει του με τον ίδιο συνεπή τρόπο που πράττουμε και εμεί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία αποδηματά, Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Äh, Κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, λυπάμαι ε, για το ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω σε όλα αυτά που είπατε και αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα υπάρξει συμφωνία ή δεν θα υπήρχε συμφωνία στο Συμβούλιο για ενισχυμένη συνεργασία. Όμως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει και μια πλειοψηφία η οποία πιστεύει ότι το σχέδιο ως έχει διαμορφωθεί δεν θα επιτύχει το στόχο που επιθυμούμε όλοι μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πρόταση ως έχει διαμορφωθεί κατά την άποψή μου δεν είναι φόρος χρηματοψητικών συναλλαγών διαρκείας, αλλά είναι περισσότερο ένα εθνικό μέτρο για να αποκτήσουν τα κράτη έσοδα, χρήματα και αυτά υπό το κάλυμα του ευρωπαϊκού φόρου. Η κυρία εισηγήτρια είπε πολύ σωστά ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να πούμε τι ακριβώς επιθυμούμε, ποια είναι η άποψή μας για την πρόταση. Πρέπει λοιπόν να πω ότι οι 11 συμφώνησαν μόνο και μόνο επειδή έκαναν ένα φοβερό τρίκ. Δηλαδή τι έκαναν. Πήραν τις δικές μας τις απόψεις επί της αρχής ότι χρειαζόμαστε αμελητή έναν φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, βιώσιμο όμως φόρο, φόρο διαρκείας και είπαν είμαστε εμείς οι 11 υπέρ του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εάν, εάν λοιπόν αυτά τα οποία θα αποδώσει θα τα εντάξουμε στον προϋπολογισμό. Ένα κομμάτι από αυτά θα τα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα μπορούμε να τα αφαιρέσουμε από τις εισφορές μας ως κράτος μέλος. Και κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να επιβάλλει αυτό το φόρο μόνο του, μεμονωμένα. Άρα δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον κοινή βάση για να υπάρξει και ένα κοινό σχέδιο. Οι μεν μιλάνε για σχέδιο Μάρσαλ, οι άλλοι μιλάνε για την καταπολέμηση της φτώχειας, οι άλλοι τη ε, ενεργείας των νέων, οι άλλοι για τους ίδιους πόρους. Έτσι λοιπόν όσο έχει διαμορφωθεί αυτή η πρόταση δεν εκπροσωπεί όλες αυτές τις απόψεις. Δεν πρόκειται να προκύψει ούτε ένα ευρώ παραπάνω στον κοινοτικό, στον ενωσιακό προπολογισμό για βιώσιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ παραπάνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που θα γίνει θα είναι να μειωθεί η εισφορά των ε, μελών. Ο δικός μου ο καγκελάριος χαίρεται διότι ανοίγει η πόρτα μέσα από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το περιθώριο που προκύπτει με αυτό το φόρο το παιχνίδι λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω το ποσοστό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να ορίσουμε ότι το ποσοστό πρέπει να παραμένει παντού το ίδιο και το ποσοστό αυτό να διοχετεύεται αναγκαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να αφαιρείται από την εισφορά των κρατών μελών. Παντού λοιπόν το ποσοστό θα πρέπει να είναι το ίδιο στα κράτη-μέλη, αλλιώς θα πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό φόρο ο οποίος θα προστίθεται στον εθνικό φόρο και με τον τρόπο αυτό θα αυξάνεται περαιτέρω ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη που θα τον εφαρμόζουν και σε εκείνα που δεν τον εφαρμόζουν. Για μένα λοιπόν αυτά που σας λέω δεν εκφράζονται επαρκώς ε, στις συμβαστικές προτάσεις. Η κυρία εισηγήτρια λέει και την καταλαβαίνω. Εμείς οι δύο τα βρίσκουμε, συνούμαστε. Δεν είναι ότι ο ένας θέλει να πονέσει τον άλλον απαραίτητα. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που είπε αυτό κατάλαβα ότι όποιος είναι υπέρ εξαιρέσεων είναι κατά του φόρου, κατά της πρώτες. Αυτό κατάλαβα. Από την άλλη όμως συμφωνούμε όλοι ότι με αυτόν τον φόρο δεν πρέπει να υπονομευτεί η ισχύουσα ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εάν λοιπόν την ρευστότητα, το αυξημένο τους αυξημένους ίδιους πόρους. Εάν δεν θέλετε αυτή τη χρηματοψητική ρύθμιση να την υπονομεύσουμε, τότε υπάρχει πρόβλημα στην ερμηνεία, διαφορετική ερμηνεία των intergroup transactions, διότι αυτές δεν είναι transactions, δεν είναι συναλλαγές, πρόκειται απλώς και μόνο για μετατοπίσεις. Γιατί λοιπόν εκφράζονται οι market makers ως εξαίρεση. Γιατί εγώ τους προτείνω ως εξαίρεση. Διότι σε πολλές χώρες οι market makers, ας πούμε Ιταλία, συγκεκριμένα Ιταλία, εκεί προβλέπεται μια ειδική ρύθμιση για τους market makers. Και εδώ η κυρία Ποδηματά έχει δίκιο. Εάν τους ε, εξαιρέσουμε αυτό θα είναι αρνητικό. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνους τους market makers που είναι ένα δυναμικό για τα μικρά χρηματιστήρια Υπάρχει λοιπόν, επηρεάζουν τα μικρά χρηματιστήρια, κατόπιν τούτου πρέπει να γίνει διαχωρισμός αυτών των market maker από το ε, εμπόριο υψηλής συχνότητας. Επ' αυτού πρέπει να συζητήσουμε. Όσον αφορά τα συνταξιωτικά ταμεία, σε τελική ανάλυση και ο Ολλανδός Υπουργός ε, Οικονομικών που αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής ε, του Eurogroup, στην ε, τελευταία κρότηση που είχε εδώ ε, σε εμά, είπε ότι η Ολλανδία δεν πρόκειται που δεν είναι να συμφωνήσει. Άρα 11 πλην 1. Δεν θα συμφωνήσει η Ολλανδία, είπε, αν τα συνταξιωτικά ταμεία λόγω της κρίσης δεν εξευρεθεί μια ειδική λύση για αυτά, μια διαφοροποιημένη. Έτσι είπε ο, ο κύριος Ντούσεμπλουμ. Άρα δηλαδή ως κοινοβούλιο εμείς δεν μπορούμε να προβούμε σε μια ρύθμιση που απλά θα οδηγεί σε ίσπραξη περισσότερων χρημάτων, χωρίς όμως να υπάρχει η ευρωπαϊκή διάσταση. Υπάρχει το ιδανικό, υπάρχει και η τρέχουσα πρόταση, ε, θα πρέπει κάπως ε, να βρεθεί μια λύση. Οι συμβιβασμοί όμως που έχουν κατατεθεί δεν αποτελούν ε, συμβιβασμού για να τους δεχθεί η δική μου η πολιτική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλώ να θυμίσω ότι η Ολλανδία δεν νίκη στους 11. Καλά. Νομίζω κυρία Ποδηματά ότι καλύτερα είναι τα σχόλια να γίνουν στο τέλος. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Το λόγο έχει ο Σερμόσα. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, είπα και στην περσμένη συνεδρίαση για το φορό των συνεργών, είναι ένας περίεργος ε, φιλελεύθερος γιατί συμφωνώ με αυτό το φόρο και δεν είναι μια θέση που συμμερίζονται και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μου. Αλλά στην τελευταία συζήτηση είπα ότι ως φιλελεύθερος φοβόμουν κάποια ανεπιθύμητα αποτελέσματα παρεμβατισμού. Επίσης μίλησα και για τις κόκκινες γραμμές μου που υπενθύμησε και ο κύριος Κάρας και γι' αυτό έχω καταθέσει τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Συμφωνώ με όσα είπε ο Ότμαρ Κάρας Δηλαδή ότι του να είμαστε υπέρ κάποιων εξαιρέσεων δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά πρέπει να εγγυηθούμε ότι τελικά δεν εμποδίζουμε την πρόσβαση χρηματοδότησης των αγορών και τελικά δεν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα όσο λειτουργούν στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές σε σχέση με τις τροπολογίες. Θέλω να πω ότι περίμενα περισσότερα από την εισηγήτρια σε σχέση με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Λάβουμε μόνο τρεις σελίδες. Θα εκτιμούσα μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερη συμφωνία με τις διάφορες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί εγώ. Θα ψήφιζα υπέρ όλων των τροπολογιών που θέλουν να εγγυθούν την δημοκρατική ποιότητα του φόρου. Θα ήμουν ε, υπέρ των τροπολογιών να ζητήσουμε από την Κομισιό να κάνει μελέτες αντικτύπου ex ante και ex post. Νομίζω ότι όλοι οι φιλελεύθεροι θα συμφωνήσουν ε, με αυτή την άποψη. Εγώ προσωπικά θα υποστηρίξω αυτές τις τροπολογίες για να εγγυηθούμε αυτό το ρόλο της Κομισιόν. Αν θα έχουμε ένα τέτοιο φόρο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι θα μπορούσε να συμβεί και τι θα έχει γίνει στις αγορές μετά από κάποιο καιρό. Επίσης, τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν ε, πρέπει να είναι μέλη της Επιτροπής του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, συμφωνώ με αυτό, και επίσης ε, θα υποστηρίξω τον ευρύτερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν βέβαια και κάποια θέματα που είναι σημαντικά για μένα και δεν έχουν επιληθεί. Όπως σας είπα, το δημόσιο ήταν κόκκινη γραμμή για μένα. Και εδώ δεν είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει ο φόρος ε, να εφαρμοστεί και στις δευτερογενείς αγορές. Και εδώ θα ήθελα είτε η συγγήτρια είτε η να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες, γιατί έχω μια ανησυχία εισαγωγή του φόρου μπορεί να κάνει τις κυβερνήσεις ακόμη πιο εξαρτημένες από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει μια τέτοια ανησυχία για ορισμένα κράτη-μέλη που εξαρτώνται πολύ από τα χρήματα της ΕΚΤ. Αν τώρα εφαρμόσουμε το φόρο και στις δευτερογενείς αγορές, μπορεί να είναι πιο εξαρτημένα τα κράτη αυτά. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν επιθυμητό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και επίσης υποστηρίζω μια τροπολογία, νομίζω ότι την κατέθεσε ο κ. Κλίνης που ζητούσε, ε, ότι το περιφερειακό χρέος ε, θα έπρεπε να χαίρει τις ίδιες μεταχείρισεις με το δημόσιο χρέος και για τα συνταξιδοτικά ταμεία. Νομίζω ότι αν δούμε την περσινή εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εξαιρεθούν τα συνταξιδοτικά ταμεία και κατά την άποψή μου οι αποταμιεύσεις ε, για τη συνταξιοδότηση ε, δεν θα πρέπει να πληρώνουν το φόρο αυτό. Επίσης, ε, θα πρέπει να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για τους market makers, τους χονδρέμπορους χρηματιστηρικών τίτλων και τις αγορές ρέπος. Γιατί ανησυχούν ε, οι αρμόδιοι από τον τομέα. Ότι αν δεν εξαιρέσουμε τους market makers και τις αγορές ρέπο, ανησυχούν μήπως ζημιώσουμε αυτές τις σημαντικούς τομείς ε, των αγορών. Εγώ θα ήμουν υπέρ λοιπόν να υπάρχουν κάποιες εξαιρεσει επί αυτών, αλλά είμαι ανοιχτό να ακούσω τα επιχειρήματα της Κομισιόν και της Ισηγητρία για να διαμορφώσω άποψη προσωπική, γιατί ξέρετε στην ομάδα μου υπάρχουν ισχυρέ απόψει επί αυτού του θέματος. Και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τη Ιταλία ε, και τη ε, Γαλλία, δηλαδή εθνική φορολογία για τα θέματα αυτά. Υπάρχει εξαίρεση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να καταβάλουν το φόρο σε εθνικό επίπεδο. Και μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης κάποιες τροπολογίες ε, που θα καταψήφιζα ξεκάθαρα όπως ε, το να κυριαρχεί η αρχή της κατοικίας. Για μένα είναι κάτι αντίθετο εδώ με την άποψη του κ. Σμιτ, δεν συμφωνώ και επίσης ε, για την εξαίρεση των παραγόγων, των hedge funds. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αντίκτυπος επί των εσόδων από αυτούς τους τομείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόσα. Εξ ονόματος των Περασίνων, ο κύριος Μπέσεκ που θα εκπροσωπήσει τον Φιλίπ Λαμπέρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι συμμερίζομαι τις απόψεις της κυρίας Ποδήματα και τις ανησυχίες της κυρίως ως προς την κρίσιμη στιγμή που ζούμε με τη συζήτηση αυτή για τον φόρο των χρηματοπιστωτικών δοσοληψιών. Είναι πολύ είναι φυσικό ότι το ξανασυζητάμε και ότι εκφράζονται και αμφιβολίες αλλά εδώ δεν πρόκειται για τεχνικές αναπροσαρμογές αλλά για να επαναλάβω τις εκφράσεις σας κυρία Ποδηματά αντιμετωπίζουμε ολόκληρη καμπάνια που στοχεύει ακριβώς την αποτυχία της εφαρμογής του φόρου αυτού. Η πίεση λοιπόν αυτή είναι ισχυρή και προέρχεται και από μερικές χώρες και από τον ίδιο το χρηματοπιστωτικό τομέα. Είδαμε ότι ο πρόεδρος της Bundesbank ο ίδιος ετάχθη κατά της αρχής της επιβολής ενός τέτοιου φόρου. Υπάρχει λοιπόν ένα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα εδώ που αντιμετωπίζουμε. Αν είναι θεμητό είναι μεν θεμητό ο χρηματοπιστωτικός τομέας να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, αν και νομίζουμε ότι υπερβάλλει πάρα πολύ τον κίνδυνο που διατρέχουν από αυτόν τον φόρο. Παρ' όλα αυτά, ο, χρηματο, ο τραπεζικός τομέας έχει στηριχθεί μαζικά και πολλές φορές έχει διασωθεί από την αλληλεγγύη της Ένωσης και των χωρών μελών. Ίσως θα έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι όλα αυτά έγιναν με τον κίνδυνο χρεοκοπίας για πολλά κράτη λόγω του κρατικού των χρέους. Και αντιμετωπίζουμε μια πολύμορφη κρίση, είναι λοιπόν φυσικό να ζητήσουμε από τον τραπεζικό τομέα που φορολογείται ιδιαίτερα χαμηλά όπως λέει και η συγγήτρια να συμμετάσχει και εκείνο στην εξέβρεση και εφαρμογή της κοινή λύσης. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τον φιλόδοξό μας στόχο, τον δικό μας και της Κομισιόν και οι συμβιβαστικές τροπολογίες και τις συμβιβαστικές τροπολογίες ιδιαίτερα δε την ιδέα που εκφράζουν αυτές ότι η φορολόγηση αυτή των δεσολυπιών θα καλύπτει το σύνολο των αγορών και των προϊόντων τους καθώς και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Το θέμα λοιπόν όπως ξαναείπα είναι κυρίως πολιτικό πια πέρα από τα τεχνικ, τις τεχνικές λεπτομέρειες του πώς και αν θα εφαρμοστεί και θα ήθελα να προσέξετε κύριοι συνάδελφοι ότι ο φόρος αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ σημαντικό και θετικό στοιχείο συμφιλίωσης των λαών με την ευρωπαϊκή ιδέα. Είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη συμβολική αλλά και πραγματική σημασία γιατί αποφέρει και κάποια χρήματα και μπροστά στις ευρωπαϊκές εκλογές που φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολες για τους θειασότες της ευρωπαϊκής ιδέας όποια και να είναι η πολιτική του τοποθέτηση δεν θα ήταν σωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση να στείλουν ένα μήνυμα που να μην στηρίζει αυτόν τον αγώνα που συζητιέται εδώ και δεκαετίες. Και τώρα για το πιο συγκεκριμένο θέμα της χρήσης του φόρου αυτού σαν, ίδιο πόρο, σαν ιδίου πόρου της κοινότητας πέρα από τις εθνικές εισφορές και όχι ως αντικατάστασή τους. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία σχετικός παρόμοια με τον κύριο Καράς και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό για να διατηρηθεί αυτός ο στόχος άκουσα αυτά που είπατε και εσείς κύριε Καράς, προτείνετε το συγκεκριμένο ποσοστό. Αλλά καταλαβαίνω και αυτό που είπατε εσείς κύριε Αποδήματα, δέχεστε την αρχή αυτής της ιδέας αλλά τονίζετε τις δυσκολίες. Είναι όμως εδώ πρόβλημα συνοχής, συνέπειας. Γιατί δεν μπορούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να έχουμε κάνει τον δημοσιονομικό αγώνα που κάναμε όλοι για να αυξηθούν οι πόροι στον προϋπολογισμό και όταν παρουσιάζεται εδώ η ευκαιρία να δημιουργεί ένας νέος ίδιος πόρος δικαιολογημένος θεμητό να υπαναχωρήσουμε. Θέλουμε λοιπόν με διατύπωση που ακόμα δεν έχει βρεθεί να διατηρηθεί αυτός ο, πόρος, ο φόρος των δοσοληψιών ως ίδιος πόρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπέσερ. Εκ μέρους ε, του ΕΣΥΑΡ, κύριο κύριος Στάσεκ. Thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούγοντας ε, τη συζήτηση για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι η εξέλιξη της στάσης, της στάσης όλων μας απέναντι στο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, των οποίων είμαι σκιώδης ηγητής επί του θέματος, εμείς λοιπόν δεν καταθέσαμε καμία τροπολογία, διότι η δική μας η θέση απέναντι στο φόρο αυτό η θέση μας παραμένει σταθερή, συνεπής, δηλαδή εμείς απορρίπτουμε αυτή την πρόταση για ουσιαστικούς λόγους και σήμερα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει και κανένας λόγος να επαναλάβουμε τους λόγους αυτούς. Πρέπει να σας πω ότι διάβασα πραγματικά πολύ προσεκτικά τις ε, σχεδόν 150 τροπολογίες και τις ε, παρατηρήσεις μου ε, τις έχω χωρίσει σε δύο μπλοκ. Στο πρώτο μπλοκ τροπολογιών, εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε, θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει. Και στο δεύτερο μπλοκ τροπολογιών διαφωνούμε. Έχουμε κάθε λόγο να τις απορρίψουμε. Ας ξεκινήσω λοιπόν με, τη, με τις τροπολογίες όπου συμφωνούμε. Συμφωνούμε λοιπόν με όλες τις τροπολογίες 21, 22, 23 και 24. Με αυτές συμφωνούμε. Αυτές είναι τροπολογίες οι οποίες οδηγούν στο να απορρίψει κανείς την πρόταση. Η δική μας στάση είναι συνεπής. υποστηρίζουμε όλες τις ε, τροπολογίες που είναι κατά αρνητικών εξωχώριων, εξωχώριες εισαγωγής του φόρου χρηματοψηφιακών συναλλαγών. Κατά τη δική μου άποψη αυτό είναι μία από τις βασικές αδυναμίες αυτού του σχεδίου. Τρίτον, εμείς ε, συμφωνούμε με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει σε μελέτη αντικτύπου και σε ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους γιατί για να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία αυτό σημαίνει περισσότερες αρμοδιότητες αλλά και δεσμεύσει από εκείνα τα κρατημέλη τα οποία δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Όσον αφορά την τελευταία ομάδα, το τελευταίο μπλοκ τροπολογιών που μπορούμε να στηρίξουμε, εμείς στηρίζουμε όλες τις απόψεις οι οποίες καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταδείξει με απόλυτη σαφήνεια ότι η εισαγωγή του φόρου αυτού δεν θα διαταράξει ούτε την κοινή αγορά, ούτε την κοινωνική συνοχή και γεωγραφική συνοχή. Τώρα πάμε σε αυτά που θα θέλουμε να απορρίψουμε. Ε, θα καταψηφίσουμε όλες εκείνες τις τροπολογίες που αντιμετωπίζουν το φόρο αυτό ως ένα εργαλείο που θα οδηγήσει στην οικονομική ανάκαμψη. Έχουμε κάνει εμπειρία με τέτοιου είδους φόρο κατά το παρελθόν και είμαστε σίγουροι ότι ο φόρος χρηματοψηφιστικών συναλλαγών θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην απασχόληση στηρίζουμε αυτές τις ε, τροπολογίες που αντιμετωπίζουν το φόρο των συναλλαγών ε, ως ε, ένα φόρο ίδιων πόρων. Υπάρχουν βέβαια και δυναμίες όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και τρίτον, εμείς είμαστε ρεαλιστές και δεν πιστεύουμε στο ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από την παγκόσμια εισαγωγή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ο φόρος σε, σε παγκόσμια κλίμακα είναι μια φρουδα ελπίδα σε επίπεδο G20. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο ε, Στάζεκ και ευχαριστούμε κύριε Στάζεκ και κυρία Ματίας εξονόματος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να έχουμε πιο αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε πριν. Εμείς, σε αντίθεση με τους συντηρητικούς, υποστηρίζουμε απόλυτα την εισαγωγή αυτού του φόρου και πρόσθετα το πρόβλημα είναι ότι έρχεται πάρα πολύ αργά και σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών. Όμως ε, δεν μπορώ παρά ότι εμείς δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει κάνει πάρα πολύ συγκεκριμένα λάθη και ευθύνεται για την κρίση που ζούμε σήμερα και δεν νομίζω ότι ένας τέτοιος φόρος θα επιδεινώσει την οικονομική κρίση. Εμεί βλέπουμε ότι η κρίση συνεχώς επιδεινώνεται αν αφήνουμε τα πράγματα και επίσης ένας από τους λόγους της επιδείνωσης είναι γιατί εμεί δεν προσδιορίζουμε, δεν λαμβάνουμε κανένα συγκεκριμένο μέτρο που να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία ρύθμιση στις χρηματαγορές και καμία παρέμβαση. Έτσι λοιπόν όλα συνεχίζουν όσοι είχαν και επιδεινώνεται η κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένω, ε, ουσιαστικά είναι πολιτικό το ζήτημα. Και εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έρχεται πάρα πολύ αργά αυτός ο φόρος. Ε, γενικά συμφωνώ με τις προτάσεις της εισηγήτριας, ε, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους. Υπάρχουν ε, κάποιες μικρές αποκλήσεις, όμως ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Θέλω όμως να κάνω κάποια σχόλια, θα ξεκινήσω από μία από τις αποκλήσεις. Εμείς ε, θεωρούμε ότι ο φόρος δεν θα πρέπει να είναι κάτω του 0,1%. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διάκριση μεταξύ του 0,01 και του 0,1. Ε, δηλαδή θα έπρεπε να είναι 0,1 για όλες ε, τις συναλλαγές και για τα ομόλογα. Γιατί βέβαια κατανοώ ότι θα είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα. Επίσης, ε, εδώ συμφωνούμε περισσότερο με την εισηγήτρια ότι ε, δεν θα θέλαμε να έχουμε μία σειρά εξαιρέσεων. Πιστεύουμε ότι όλες οι χρηματαγορές και όλα τα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται ειδικά όταν μιλάμε για ε, κάποιες συναλλαγές με κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όχι, ε, μας δεν μας ενδιαφέρει να γίνεται αυτή η διάκριση. Πιστεύουμε ότι όλα θα πρέπει να καλύπτονται από το φόρο. Και αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, αν ε, έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται κάτι ακόμη για να υποστηρίξω την πρόταση ο φόρος αυτός να χρησιμεύσει για να ενισχύσει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως ήδη ε, πόρη. Αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί παρά να έχει δική του θέση για το θέμα αυτό. Και εγώ νομίζω η θέση μας πρέπει να είναι η ενίσχυση του προϋπολογισμού. Και να πω και πάλι ότι εμείς ε, δεν μπορούμε να αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση του προπολογισμού, την αύξηση των κονδυλίων ε, στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και κατόπιν να υποστηρίξουμε ένα μέτρο που θα μειώσει τις συνεισφορές των κρατών ε, στα πλαίσια του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έτσι λοιπόν νομίζουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όσοι διπόρεις θα μπορούσε να φτάσουμε στα 30 και πάνω από τα 30 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και φυσικά πρέπει ε, να δούμε ε, και πώς θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας ε, και ανάπτυξη κάτι ακόμη για να αναφερθώ σε κάτι που δεν συζητήθηκε εδώ και έχει να κάνει με τη φορολόγηση. Εγώ παρουσίασα κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε κοινά μέτρα που να, απο, να, να καταπολεμούν την φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη και στο πλαίσιο αυτό. Δεν συμφωνώ με τη θέση να αφήσουμε σε κάθε κράτος μέλος να προσδιορίσει τα μέτρα αυτά για την πρόληψη της ε, φοροδιαφυγής και της φοροποφυγής για ένα πολύ απλό λόγο. Εμείς ξέρουμε ότι αν τα αφήσουμε αυτά στα κράτη-μέλη δεν θα γίνει τίποτα ή πολύ λίγα. Έτσι λοιπόν ε, χρειαζόμαστε μια κοινή δράση που να μας επιτρέψει να γίνει μια διαρθρωμένη παρέμβαση. Διαφορετικά φοβάμαι ότι πάρα πολύ λίγα θα γίνουν και για μια ακόμη φορά δεν θα αποφύγουμε αυτή την ε, συνήθη πρακτική. Δηλαδή φοροδιαφυγή. Και αν ε, δούμε κάποια παραδείγματα, αρκεί να δούμε τι έγινε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. βλέπουμε ότι όταν χρειάζονται ε, να αναλυφθούν μέτρα, τίποτα δεν γίνεται, γι' αυτό πρέπει να αναλυφθεί κοινή δράση. Λεχθέντος αυτού. Συμφωνώ με τις περισσότερες από τις προτάσεις της εισηγήτριας και θα την υποστηρίξουμε στο επίπεδο αυτό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Ματίας. Γκοσές, Λούλινγκ, Κλίντ, Σμιτ, Φερέιρα, Γκαιόν και Φέρμπερ έχουν ζητήσει το λόγο. Αν κάποιος άλλος ε, θέλει το λόγο να μα το πει τώρα. Καταρχήν ο κύριος Γκοσές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Καταρχήν δέχομαι αυτά που είπε ο συνάδελφος Καράς και επί των αρχών και επί των τεχνικών προβλημάτων. Πρέπει όμως σήμερα να αναρωτηθούμε το εξής. Μήπως δεν υπαναχωρούμε επί της αρχής του φόρου αυτού. Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για υπαναχώρηση, αλλά για μια ρεαλιστική εξέταση. Όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια φορολογία δεν υποκύπτουμε ούτε σε ηθικές αρχές ούτε σε ρομαντισμούς γιατί ο στόχος της φορολόγησης είναι να πάρουν τα κράτη-μέλη και οι δημόσιοι οργανισμοί τα έσοδα που χρειάζονται για να καλύψουν τις δαπάνες τους. Ζητούμε λοιπόν και αποτελεσματικότητα και πραγματισμό, ρεαλισμό. Βλέπουμε όμως ότι όσο πιο κοντά βλέπουμε τους αριθμούς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν είχαν από την αρχή προβλεφθεί ούτε από την Κομισιόν ούτε από άλλους. Η αρχή της φορολόγησης αυτή ήταν απλή και αρκετά ικανοποιητική. Λέγαμε δηλαδή ότι θα φορολογηθούν οι διάφορες δοσοληψίες, αυτό θα καταλήξει και σε περισσότερο ηθικές δοσοληψίες, πόσο μάλλον που ο φόρος θα είναι πολύ χαμηλός. Επ' αυτού συμφώνησε μεγάλη πλειοψηφία και στήριξε την αρχή αυτή. Σήμερα όμως το θέμα είναι όταν βλέπουμε τις λεπτομέρειες μήπως αυτά που κάνουμε δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν δηλαδή. Να μην είναι τιμωρητικός ο φόρος αυτός λέγοντας ο χρηματοπιστωτικός τομέας έκανε το α και το β πρέπει να τιμωρηθεί. Το θέμα δεν είναι να τιμωρηθεί σήμερα είναι να μην έκανε αυτά που είχε κάνει πριν που δεν αλλάζουν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να είμαστε τιμωρητικοί. Δεύτερον, είναι χήμερα να πούμε ότι θα βελτιωθεί έτσι η χρηματοδότηση της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη μάλλον θα αποζητήσουν περισσότερους πόρους για τους εαυτούς τους, δηλαδή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μεσοπρόθεσμα δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Άρα το θέμα είναι πώς η φορολόγηση αυτή θα έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Γιατί προοδευτικά αν καταλήξει να καταστρέψει τις οικονομικές δραστηριότητες ή να υπάρξει διαφυγή θα είναι κάτι αρνητικό αν βασίζεται σε κάτι που λόγω ακριβώς των στρεβλωμένων δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτό ζητούμε στο Κοινοβούλιο έναν ικανοποιητικό και αποδεκτό συμβιβασμό. Χρειάζεται λοιπόν πολύ ακόμα δουλειά, αλλά επίσης όσοι επικρίνουν το φόρο αυτόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμπάνια εναντίον του φόρου, το είπα και στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα, είναι φυσικό ο φορολογούμενος να ζητάει να πληρώνει όσο το δυνατόν λιγότερα το κράτος πρέπει να το φροντίζει αυτό για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Αλλά πρέπει και οι μέλλοντες φορολογούμενοι να μην περιορίζονται στα λόγια μόνο. Και γι' αυτό ζητάω και από τους μεν και από τους δε τους επικριτές του φόρου να μας δώσουν αριθμούς που να επιτρέπουν να μετρήσουμε τις πιθανές ζημίες που θα προέλθουν από αυτήν τη φορολόγηση, τη διπλή φορολόγηση κλπ αριθμούς δηλαδή που ακούγονται αλλά επί των οποίων δεν θα μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι παρά μόνο αν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς. Μέχρι σήμερα υπάρχει μεγάλος δισταγμός για την αναφορά τέτοιων συγκεκριμένων δημοσιονομικών στοιχείων και αριθμών. Χωρίς αυτούς όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε θέσεις αξιόπιστα. Γι' αυτό λέω έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Βέβαια είναι συμβουλευτικός ο ρόλος μας αλλά δεν είναι αυτό αιτία για να λέμε ότι μας κατέβει. Τα κράτη ούτως ή άλλως θα κάνουν ό,τι θέλουν και εμείς πρέπει να φροντίσουμε η συζήτηση να είναι κατανοητή από τους πολίτες, δίκαια για την οικονομία και να κινείται προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και όχι σε μείωση της δραστηριότητας μέσω του, της χρεοκοπίας επιχειρήσεων που μπορεί και αυτές να δικαιολογούνται αλλά όχι πάντοτε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ διαπιστώνω με μεγάλη ευχαρίστηση ότι στις συζητήσεις μας Υπάρχει τώρα πιο πολύς ρεαλισμός. Ξέρω ότι δεν είναι πια η εποχή της συζήτησης του κατά πόσον είναι θεμητός ο φόρος αυτός. Αυτό, η συζήτηση αυτή έχει ήδη γίνει και πολλές φορές. Θέλω όμως να παρατηρήσω γενικά ότι ο φόρος αυτός, το έχω ξαναπεί, φαίνεται ότι κάθε μέρα συναντάει και καινούργιες δυσκολίες και ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακόμη κι αν κανείς είναι αναφανθόν υπέρ αυτού του φόρου, πρέπει να αναγνωρίσει τις δυσκολίες και όχι να τις αρνείται. Γιατί ορισμένοι φαίνεται ότι είναι τυφλωμένοι και δεν βλέπουν τα πράγματα όπως είναι και αυτό δεν βοηθάει την επίλυση του προβλήματος ενός φόρου που υποτίθεται ότι θα καταπολεμήσει και δικαίως τις τρευλώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά που τελικά μπορεί να καταλήξει στο να πληρώσουν την ύφη οι καταναλωτές. Γιατί θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι θα τιμωρηθούν οι χρηματοπιστωτές, οι καταναλωτές εκείνοι που αγοράζουν τις υπηρεσίες θα τιμωρηθούν. Όσο για... Όσο για την ετεροδικία, δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι πρόκειται σαν ένα είδος ενισχυμένης συνεργασίας που θα υποχρεώσει τελικά όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το φόρο αυτόν και ότι τάχα αυτό δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ή δεν θα θέσει δυσκολίες. Δεν λέω ότι αποκλείεται η εφαρμογή, ότι δεν γίνεται, αλλά η κοινότητα των νομομαθών ε, έχει πολλές αμφιβολίες και το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε την προσφυγή του για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις τώρα εγώ προσωπικά πάντα είχα αμφιβολίες αλλά δεν είμαι και ταγμένη κατά αναφανδών τουλάχιστον ο τρόπος εφαρμογής όμως του φόρου αυτού όπως έχει αναλυθεί μέχρι τώρα δεν με ικανοποιεί και γι' αυτό έχω καταθέσει ορισμένες τροπολογίες. Το θέμα των συνταξιοδοτικών ταμείων και χαίρομαι γιατί και άλλοι συνάδελφοι κατέθεσαν ανάλογες τροπολογίες και των επενδυτικών ταμείων είναι ουσιώδη θέματα. Είναι κόκκινη γραμμή για μένα και για άλλους. Αν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία δεν αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του φόρου αυτού, τότε εγώ θα καταψηφίσω. Γιατί μερικοί δεν γνωρίζουν ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι από τον φόρο αυτόν σε βαθμό που μπορεί να χρεοκοπήσουν ορισμένα ταμεία αναπήρων κλπ. Δυστυχώς από ιδεολογική προκατάληψη η Κομισιόν δεν θέλησε ποτέ να αναγνωρίσει ότι η φορολόγηση τέτοιων ταμείων θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για αυτά. 10, 20, 30 φορές αν εφαρμοστεί ο νόμος αυτός του 0,1% θα οδηγούσε σε απαγορευτικά ποσοστά και δεν καταλαβαίνω ότι ούτε καν το αναγνωρίζουν αυτό το πρόβλημα. Είναι παράλογο διότι έτσι τιμωρούμε την αποταμίευση και τα όργανα συλλογής αποταμίευσης που είναι σταθεροποιητικοί παράγοντες. Εξάλλου και τα οσεκά θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε χωρίς να χρειαστεί να πάμε στη Σιγκαπούρη κλπ. Θέλετε να εφαρμοστεί ένας νόμος για να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία, αλλά αν καταλήξουμε να τιμωρήσουμε έτσι τα εργαλεία συλλογή της αποταμίευσης, νομίζω ότι διανοητικά υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτόν τον συλλογισμό και τον οποίο εγώ καταδικάζω στεναρά θα ήθελα να ακούσω και τους άλλους, ορισμένους τους έχω ακούσει, που έχουν παρόμοιες αντιρρήσεις, αλλά φυσικά αυτό το θέμα είναι για μένα καθοριστικό και δεν μπορούμε να παραλείψουμε μία εις βάθος εξέταση του. Η κυρία Σιγήτρια είπε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Εγώ δεν έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω αν είναι αισιόδοξη ίσως και ουτοπίστρια. Αλλά δεν έχω δει ακόμη τις συμβιβαστικές τροπολογίες από τους κοιόδης. Θα κάνω και εγώ ό,τι προσπάθεια γίνεται για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς, ελογικούς συμβιβασμούς. Αλλά από ό,τι άκουσα μέχρι τώρα από την εισηγήτρια και όσους την υποστηρίζουν δεν με έχει πείσει. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω να κάθεται εδώ ο κύριος Μπέρκμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω την υπομονή του και τον, την ιδεολογία του. Γιατί η πρόταση την οποία κατέθεσε και που είναι το σημείο κίνησης συζήτησης, εντωμεταξύ διαφοροποιείται πάρα πολύ από εκείνο το οποίο συζητάμε εμείς τώρα. Έκανε λοιπόν ένα πολύ θαραλέο βήμα και πρότεινε κάτι που αν το είχαμε εφαρμόσει πράγματι ε, θα είχε τη δυνατότητα να έχει παγκόσμιε προεκτάσει. Αυτά που συζητάμε σήμερα δεν έχουν πια πολλά κοινά στοιχεία με την αρχική πρόταση. Και δεν θα εκπλαγώ αν ο κύριος ε, Μπέρκμαν είπε φτάνει πια, εγώ ε, ξέρουμε δεν ενδιαφέρομαι πια. Κοιτάξτε, ο φόρος έχει δύο στόχους. Αφενός έχει ε, το στόχο τη ρύθμιση των πραγμάτων και αφετέρου έχει ω στόχο ένα φόρο να φέρει χρήματα στον κορβανά. Αυτή ήταν και η αρχική ρύθμιση. Εγώ νομίζω από την πρώτη αρχή τα περί της ρύθμισης αποστασιοποιηθήκαμε πάρα πολύ και παραμείναμε στο δεύτερο του πώς θα φέρουμε περισσότερα χρήματα στον ενωσιακό κορβανά. Ε, λένε περικοί ότι είναι πρόθυμοι να εισάγουν τον φόρο αυτό ε, λέγεται αυτό. Το να πιστεύει όμως κανείς ότι αυτό θα το κάνει από μόνος του ο χρηματοψηφιστικός τομέας, αυτό είναι πλάνη. Ε, σε τελική ανάλυση θα ε, μετακυλιστούν αυτά τα χρήματα στους, ε, τραπεζικούς, ε, στους πελάτες των τραπεζών. Αυτό που είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι και οι 11 δεν συμφωνούν ούτε τι θέλουν ούτε πώς θα επιδιώξουν αυτό που επιθυμούν. Ας δούμε λιγάκι τα πράγματα πρακτικά. Έχουμε 11 υπουργού οικονομικών οι οποίοι συζητάνε γι' αυτό το, το φόρο. Ο Λανδός λέει εξαιρούνται τα συνταξιωτικά ταμεία. Ο Βρετανός λέει εξαιρούνται τα ΟΣΕΚΑ. Ο Γερμανός ε, λέει η σύνταξη Ρίστερ ε, Ξέρετε και αυτή. Οι Γάλλοι λένε μα τον φόρο αυτό τον εισαγάγαμε εμείς το καλοκαίρι και δεν χρειάζεται να εφαρμόσουμε τίποτα. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε μιλάμε για τον πύργο της Βαβέλ. Ε, τέτοιου είδου συνθήκες όταν μιλάνε οι Υπουργοί Οικονομικών για το φόρο χρηματοψηφιακών συναλλαγών. Ο κ. Μπέρκμαν είχε δώσει έναν ορισμό, εντωμεταξύ όμως ε, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά πράγματα κατά νου. Πέρα από αυτό λοιπόν δεν συμφωνεί κανείς με αν τελικά προκύψουν χρήματα από το φόρο αυτό, τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά. Οι μεν λένε θα μπουν στον προπολογισμό ο δικός μου ας πούμε Υπουργός Οικονομικών της δικής μου της χώρας ε, μιλάει ήδη για δύο δις ε, πλασματικά αυτή τη στιγμή αλλά τα εντάσσει τον προπολογισμό ως μελλοντικά έσοδα. Ίσως το ίδιο να έκαναν και άλλοι. Άλλοι πάλι να λένε ότι το σύνολο των εσόδων θα διοχετευτεί στον ενωσιακό προεπολισμό θα μειωθεί βέβαια αντίστοιχα η εθνική συνεισφορά. Βλέπετε λοιπόν υπάρχει τεράστια δυσαρμονία ε, σε αυτά που λέγονται. Εγώ τολμώ να πω δεν θα επιβληθεί ο φόρος αυτός άσχετα με το τι θα συζητάμε εδώ. Σε τελική ανάλυση οι 11 δεν θα συμφωνήσουν. Βέβαια δεν αποκλείω να έρθουν ε, κάποιες ε, σπασμωδικές ε, φορολογήσεις στις, με τα, στις συναλλαγές μετοχών, ένα είδος stamp duty του φόρου του χαρτοσύμου. Επειδή λοιπόν πιστεύω ότι τελικά ένας φόρος που προκαλεί στρεβλώσεις δεν είναι σκόπιμος, γι' αυτό και εγώ προτείνω όλα αυτά να τα εισάγουμε σταδιακά. Να ξεκινήσουμε δηλαδή με κάτι με το οποίο συμφωνούν και 27, σύντομα 28. Ένα είδος φόρου χαρτοσύμου, όπως το έχουν οι, οι Άγγλοι. Με αυτό να ξεκινήσουμε και αν λειτουργήσει μετά από 2-3 χρόνια ε, σταδιακά να αυξήσουμε το φόρο. Αυτά όμως που λέμε τώρα φοβάμαι ότι θα αποτύχουν ικτρά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σμίθ έχει τώρα το λόγο. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους είπαν κάτι σαν στο έλεγα. Δεν μου αρέσουν αυτά τα σχόλια, αλλά δυστυχώς τώρα νομίζω πρέπει να το κάνω. Θα έλεγα κάπως διστακτικά το πράτο. Αλλά φυσικά αυτό συμβαίνει αν μπει στις λεπτομέρειες και αν μελετήσει τις λεπτομέρειες και προσπαθήσει να καταλάβει αυτά που είπε και ο φίλος μου είπε ότι θέλει το φόρο από τον κύριο Μπέρκμαν αλλά όχι αυτό το φόρο και δεν θέλει τις εξαιρέσεις λοιπά. Μήπως ε, θα πρέπει να την αφήσουμε κατά μέρου στην όλη και να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Η ιδέα του να έχουμε ένα φόρο για την πρόθεση της ανάπτυξης στην Ευρώπη μπορεί και να μην είναι τόσο εξαιρετική. Δεν ξέρω. Έχουμε αυτές τις εμπειρίες ε, στην πατρίδα μας ε, και δεν μπορούν να συγκριθούν. Συμφωνώ εν μέρη, αλλά Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες σε λεπτομέρειες. Ε, άκουσα τι είπε ο κύριος Γκίγκολ ότι οι χώρες που είναι εκτός ε, δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο ή τουλάχιστον ισχυρό λόγο. Πάντοτε πολύ βγαίνει βέβαια τα λέτε αυτά, δεν σας ασκώ κριτική, όμως προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αν ε, αυτό το κλαμπ των 11 προχωρήσει. Μήπως ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι δυνατό να μην επηρεάσει και τις υπόλοιπες χώρες που είναι εκτός με τις συνθήκες που έχουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εξοδαφικές πτυχές δεν έχουν εξεταστεί πλήρως. Και δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. τουλάχιστον για αυτές τις χώρες ε, που δεν συμμετέχουν στο μηχανισμό, σε αυτόν τον κλαπ των 11, θα μπορούσε να είναι κάτι αποδεκτό αυτό. Και κλείνοντας θα έλεγα... Εσείς που θέλετε αυτό το φόρο, θα έπρεπε τελικά να πείτε αν ε, εδώ στοχεύεται στα έσοδα για να προκείται για πολιτικό συμβολισμό. Εγώ συμφωνώ ότι οι χρηματαγορές πρέπει να ρυθμιστούν με πιο αυστηρό τρόπο. Ακόμη και εγώ μπορώ να το δεκτώ αυτό. Αλλά αν εισαγάγουμε ένα τέτοιο φόρο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και θα πρέπει και να κατανοηθεί σε ευρύτερη προοπτική. Έτσι λοιπόν ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν θα έλεγα καλή τύχη ή bon sens, γιατί θα το καταψηφίσω όπως και να έχει. Αλλά καλή τύχη στην εισηγήτρια, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Muchas gracias. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σμιτ. Η κυρία Σας ευχαριστώ. Έχω χαθεί κάπως με τα επιχειρήματα που ακούγονται. Γιατί Ακούμε το επιχείρημα ότι θα πληρώσουν οι καταναλωτέ. Ναι, αυτό είναι ένα μέρος του επιχειρήματος ε, που υιοθετώ. Όμως, σας παρακαλώ να θυμάστε ότι οι καταναλωτές ακόμη και για ένα βιβλίο στη χώρα μου πληρώνουν 23% ΦΠΑ. Γιατί αν παραδείγματο χάρη, αν δεν αγοράζουν ένα βιβλίο ε, ή ένα μπουκάλι νερό αγοράζουν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν. Επίσης, να μιλήσουμε για την αντίληψη των πολιτών πληρώνουν πάρα πολλά οι πολίτες και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Καταβάλουν πάρα πολλά στο διεθνή, στον εθνικό προϋπολογισμό και έμεσα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και αυτή η απαλλαγή του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι πάρα πολύ μικρή όταν τη συγκρίνουμε με την πραγματική οικονομία. Δηλαδή θα έπρεπε οι καταναλωτέ και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα να πληρώνουν και αν και ο χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να πληρώσει περισσότερο και αυτό είναι εντάξει. Αυτό. Τώρα να μιλήσουμε για τι εξαιρεσει. Λυπάμαι, αλλά δεν ε, καταλαβαίνω γιατί προτείνεται να εξαιρεθούν τα συντοξιδωτικά ταμεία. Δεν είναι μικρές επιχειρήσει, είναι μεγάλε επιχειρήσει. Δεν ε, θα καταστραφούν και επειδή θα πρέπει να πληρώνουν το 0,1% φόρο επί των συναλλαγών του. Αυτό θα γίνει μόνο αν επενδύουν σε πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα με μεγάλη επιθετικότητα και σε συναλλαγές υψηλή συχνότητας. Μόνο τότε θα θυγούν από αυτό το φόρο. Αλλά αυτή είναι μια θετική συνέπεια γιατί τα συνδοξιδωτικά ταμεία θα έπρεπε να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα και όχι σε βραχυπρόθεσμα προϊόντα. Και το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο χρέος. Γιατί το δημόσιο χρέος βγήκε εκτός ελέγχου όχι επειδή υπήρχε επανάπτυξη, αλλά επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη κερδοσκοπία στην αγροπολισία δημοσίου χρέους και CDS. Και γι' αυτό αυτό οι αγορές τώρα είναι πιο σταθερές μόνο επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άρχισε να υλοποιεί τις νομισματικές συνελλαγές. Γιατί στο παρελθόν, όταν υπήρχε κερδοσκοπία, ήταν πολύ ψηλό και το χρέος. Ας μην τα μπερδεύουμε λοιπόν όλα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν καλή λόγια για όλες τις εξαιρέσεις. Ε, τώρα, για τις ε, τροπολογίες. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σοβαρά, αλλά ας δούμε τι έχουν προτείνει οι διάφοροι συνάδελφοι ως εξαιρέσεις από το φόρο. Τις ε, ενδομιλικές ε, συναλλαγές, δεν θα αναφέρω τώρα τις τροπολογίες, και τις συναλλαγές μεταξύ ομίλων ε, όταν πληρούνται οι απαιτήσει προστασίας και θέλουν να εξαιρέσουν την επαναγορά της συμφωνίες δανεδότησης και δανεισμού. Άλλη ομάδα βουλευτών θέλει εξαίρεση για τους ΟΣΕΚΑ και εναλλακτικά ταμεία επενδύσεων. Άλλοι θέλουν να τα συντοξιδοτικά ταμεία ε, να εξαιρεθούν. Ε, άλλη ομάδα θέλει να εξαιρεθούν τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να εξαιρεθούν τα εξωχρηματιστηρικά προϊόντα και η δραστηριότητα των χονδρέμπονων χρηματιστηρικών συναλλαγών, εξαίρεση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εξαίρεση για τα μέσα που εκδίδονται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξαίρεση των υποκατεστημάτων που έχουν έδρα σε ένα συμμετέχον κρατομέλος αλλά λειτουργούν σε ένα μη συμμετέχον κρατομέλος όταν ε, δεν υπάρχει εμπορία σε μέσο που εκδίδεται από συμμετέχον κρατομέλος. Εξαίρεση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, εξαίρεση μέσων που εκδίδονται από μη συμμετέχοντα κράτη-μέλη, εξαίρεση του δημοσίου χρέους, εξαίρεση των ε, παραγών που σχετίζονται με τα επιτόκια, εξαίρεση για τα ομόλογα, την πρωτογενή αγορά, για τις επιχειρήσεις σε παράγωγα και άλλα. Για να σας ρωτήσω λοιπόν δεν είναι αυτή μια στρατηγική να αποδυναμωθεί εντελώ ο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσω των εξαιρέσεων. Εγώ μπορώ να βρω πάρα πολλού λόγου να εξαιρέσουμε, αλλά εδώ τι θέλουμε να καταπληκτήσουμε, τι είναι υπερβολική εμπορία χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Είστε σίγουροι ότι όλοι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, ότι ω εκπρόσωποι των πολιτών μπορούμε να προχωρήσουμε με μία θέση να ανοίξουμε δηλαδή όλα αυτά τα νομικά κενά. Και φυσικά ε, έχουμε πολλούς λόγους να τα ξερέσουμε όλα αυτά αν δεν λάβουμε υπόψη τη γενική εικόνα, αλλά σας παρακαλώ ας είμαστε σαφείς και ειλικρινείς. Και σε ό,τι αφορά τις κατοχώρες, εγώ ξεπλάγει, δεν είναι μία από τους 11 η χώρα αυτή, είναι εκτός. Είστε λοιπόν κύριε Κάρας, είστε σίγουρος ότι αν αποκλείσουμε τα τα ταμεία, οι κάτω χώρες σας συμμετέχουν. Ε, δεν το νομίζω. Γιατί. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Είπε κάποια πράγματα σαφή, ότι ένας από τους λόγους που ήταν εκτός ήταν τα τα ταμεία. Δεν είπε όμως ότι αν εξαιρεθούν αυτά θα συμμετέχει η Ολλανδία. Ας είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε μια κοινή θέση από το Κοινοβούλιο, εδώ δεν μιλάμε για συναπόφαση θα πρέπει να μείνουμε στην αρχική μας θέση, δεν θα έπρεπε να ανοίξουμε παραθυράκια, γιατί τελικά όλα αυτά θα γίνουν μεγάλες ορθάνυχτες πόρτες για τις εξαιρέσεις και θα καταστρέψουν τελείως το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτή είναι η θέση μου. Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Ο κύριος Γκίκολ. Well, uh, like to... Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίσα που είπε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και εγώ αλλά τα είπε με καλύτερο τρόπο από ό,τι θα τα έλεγα. Την ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Δεν θα επισέλθω σε καμία από τις συγκεκριμένες προτάσεις αλλά έχω και εγώ την ίδια εντύπωση. Ξέραμε βέβαια από πολύ καιρό ότι είναι αμφιλεγόμενο το θέμα από τότε που το πρότεινε ο Κέινς. Επομένως, Ραμόν, μην εκνευρίζεσαι που είσαι φιλελεύθερος και υπέρ του φόρου. Και ο Τζον Μέιναρτ Κέινς φιλελεύθερος ήταν από τη δική σας ιδεολογική οικογένεια όταν το πρότεινε. Αλλά βέβαια φιλελευθερισμός είναι, ο φιλελευθερισμός παραβιάζεται όταν ασχολούμαστε μόνο με τη φορολόγηση ορισμένων προϊόντων και όχι άλλων. Διότι τότε δεν ακολουθούμε ισότιμη μεταχείριση που είναι η κύρια ιδέα μιας κοινωνικής αγοράς ε, και μιας σωστά διευθετημένης αγοράς. Υπήρξε λοιπόν μακρά συζήτηση και διαφορές και είναι ενδιαφέρον ότι έχουν αλλάξει στάση ορισμένοι γιατί μερικοί, από ήταν κατά, μερικοί κατάλαβαν ότι δεν είναι και τόσο κακή ιδέα άλλοι πιστεύουν ακόμη ότι μπορούν να σταματήσουν την εφαρμογή του φόρου και ζητούν πιο ενδιαφέρουσες, πιο έξυπνες μελέτες να ανοιχθούν κατά του φόρου και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα που είναι η πιο επικίνδυνη μέχρι τώρα. Αυτοί κατάλαβαν τον αρχή «If you can't beat them, join them». Και γι' αυτό λένε ότι και αυτοί υποστηρίζουν το φόρο αλλά προσπαθούν να τον υπονομεύσουν από τα μέσα με πολλούς τρόπους όπως ένα μακρύ κατάλογο εξαιρέσεων και μια άλλη στρατηγική είναι να επιμηκυνθεί η όλη διαδικασία παρεμβάσεων και το πιο επικίνδυνο από όλα, η πιο επικίνδυνη από όλους είναι εκείνοι που δεν δείχνουν τα επενδεδημένα συμφέροντά τους. Εγώ ανησύχησα όταν η ΕΚΤ είπε ότι καταρχάς είναι κατά του φόρου αλλά τώρα δημόσια λένε ότι θέλουν και αυτοί να γνωμοδοτήσουν. Δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να ζητούμε συμβουλές από ανθρώπους που δεν υποστηρίζουν κάποια ιδέα. Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα και μόνο μία δικαιολόγηση υπάρχει για τις εξαιρέσεις. Η περίπτωση όπου δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τη φοροδιαφυγή με βάση ένα από αυτά τα προϊόντα που φορολογεί ή αφόσον βέβαια έχει ήδη χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα νομικά μέσα. Αν δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή τότε φτάνει στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Σουήδοι. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Αλλά πέρα από αυτό όλες οι προτάσεις που λένε ότι αφού είναι καλό πράγμα οι συντάξεις να μην φορολογούνται ε, και για αυτές χρησιμοποιούνται καμιά φορά λένε οι φοροαπαλλαγές και φοροδιαφύγες όχι όλα αυτά στοχεύουν στην καταστροφή της ισονομίας και τελικά υπονομεύουν την όλη ιδέα του φόρου και βέβαια τμήμα του φόρου φυσικά θα πληρωθεί και από τους χρήστες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν είναι και αυτό κακό πράγμα εφόσον όλοι θα χρησιμοποιούν ισότιμα, θα φορολογούνται ισότιμα από τέτοιου είδους υπηρεσίες. Και τέλος αυτά που είπε ο Όλε. Είδα τις τροπολογίες ορισμένων συναδέλφων που ζητούν συνολική απόρριψη. Αν συνδυάσουμε τις δικαιολογήσεις και του Όλε και του Γκούναρ Χόκμαρκ και ορισμένων άλλων από το ΕΛΚ πρέπει να ομολογήσει ότι είναι περίεργες διότι η απόρριψη της πρότασης εφόσον βασίζεται σε ενισχυμένη πλειοψηφία θα σημαίνει ότι θεωρείται ότι έχει πολύ αρνητικές συνέπειες σε χώρες που δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή του φόρου. Προτείνονται δηλαδή από ευρωβουλευτές που, από χώρες που δεν έχουν ενταχθεί στην ιδέα αυτή. Άρα τι νόημα έχουν όλα αυτά. Οι χώρες που συνεργάζονται έχουμε αναρωτηθεί ήδη πρέπει να είναι οι μόνες που θα γνωμοδοτήσουν ή και οι υπόλοιπε. Δεν θελήσαμε να κάνουμε υποδιαιρέσεις, μια υποεπιτροπή δηλαδή με διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα με το αν κανεί στην Ευρωζώνη ή όχι, αλλά παρόλα αυτά αμφισβητείτε εδώ το κατά πόσον όλα αυτά είναι θεμητά. Πρέπει όλοι μαζί να αναλάβουμε την ευθύνη. Και στο Συμβούλιο υπάρχει ο κίνδυνος χώρες που δεν έχουν καμία πρόθεση να ενταχθούν να διαταράζουν τη διαδικασία. Και εδώ θα μας ρωτήσουν αργά ή γρήγορα γιατί συζητούμε όλοι μαζί αυτά τα πράγματα. Ενώ ορισμένοι με τα κόμματα που εκπροσωπούν καταπολεμούν τον φόρο και δεν πρόκειται να τον εφαρμόσουν. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι νομικό επιχείρημα, αλλά το θέμα είναι τι και πώς θα χειριστούμε το θέμα ώστε το Κοινοβούλιο να φανεί ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι όλοι τα μέλη του από χώρες της Ευρωζώνης είναι το Κοινοβούλιο του Ευρώ. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πώς θα δικαιολογήσουμε όλες μας τις προτάσεις και τροπολογίες. Αυτά τα ερωτήματα τίθενται και θα τεθούν και είναι σωστό να τεθούν. Ο κύριος Φάρμπερ τώρα. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρέπει να σας πω ότι λυπάμαι λιγάκι για το γεγονός ότι την πρότασή μου θα την απορρίψουν οι σοσιαλιστές. Γιατί βασικά είχαμε συμφωνήσει και με μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία να ταχθούμε υπέρ του φόρου ε, χρηματοψηφιτικών συναλλαγών. Και τώρα καλούμεθα στο σκελετό να δώσουμε σάρκα και οστά. Εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι από τη Μία πλευρά υπάρχουν οι μεν που λένε ότι ορισμένα παράγωγα ε, δεν θα πρέπει να φορολογούνται και τα ίδια παράγωγα όμως ε, στην περίπτωση που πρόκειται για υπέρμετρη κερδοσκοπία, αυτά να φορολογούνται. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω με απόλυτη σαφήνεια ότι η τροπολογία την οποία κατέθεσα, η τροπολογία αυτή φύγει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, εκεί όπου ως ε, Ήπειρος, με ουσιαστική παραγωγή. Επιθυμούμε να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα την παραγωγή μας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ήχου, κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν παράστα, παρεμβολές, κάτι δεν πάει καλά. Σταματάει και ο μιλητής. Λοιπόν, συνεχίζει. Ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς που υποφέρουν, λέει ο μιλητής. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Λοιπόν, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι δυνατόν να προκύπτει υπεραξία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να απευθυνθώ κυρίως στους συναδέλφους τους σοσιαλιστές και να τους πω ότι αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει αλλού να τα συμπεριλάβουμε και εδώ, στο φόρο χρηματοψηφιωτικών συναλλαγών. Ε, θα ήθελα να φερθώ στο τελευταίο θέμα που είπε και ο κύριος Γκίγκολτ, γιατί αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εντωμεταξύ έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποτελεί από διάφορα τμήματα. Εμείς ως Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα ως Οικονομική Νομισματική Επιτροπή εκπροσωπούμε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 και σύντομα τους 28. Έχουμε κατόπιν την Ένωση ε, των 25 έχουμε κατόπιν ε, τους 17 την Ευρωζώνη και τώρα θα έχουμε και την Ένωση των χωρών που θα εισάγουν το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τις 11 αυτές ε, χώρες. Όπου λοιπόν δεν είμαστε 27, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλά παριστάμεθα ως ακροατές, είμαστε ιδιαίτερα αδύναμοι. Γι' αυτό λοιπόν για μας ε, είναι όλο και πιο δύσκολο να ε, μεταφέρουμε τις απόψεις μας προς τους απλούς πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν με σαφήνεια αυτό το διαχωρισμό των 11, των 25, των 27 ε, αντιμετωπίζουμε λοιπόν πρόβλημα και γι' αυτό θέλω να σας πω με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτοί οι οποίοι είπαν ότι δεν θα ενταχθούν στους 11 αυτοί δεν μπορούν να λένε ότι εμάς δεν μας αρέσει, δεν θα εισαχθεί ο φόρος αυτός. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της ενισχυμένης συνεργασίας και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εμείς ως Κοινοβούλιο να τοποθετηθούμε που δεν θα είναι απλά ένα τυπολατρικό στοιχείο, δηλαδή κάναμε μια γνωμοδότηση, αλλά να ακολουθήσει και νομοθετική διαδικασία. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, στο μέλλον δεν θα παίζουμε κανένα απολύτως ρόλο. Και αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι σε τελική ανάλυση υπάρχει ο κίνδυνος ε, να υποστούμε την κατάτμιση της ε, Ευρώπης, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για τους πολίτες της Ευρώπης. Ο κύριος Λάγκεν. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι σύντομος. Τα περισσότερα επιχειρήματα τα οποία ήθελα να φέρω αναφέρθηκαν και επιθυμώ να αναφερθώ στην πλήρη εξαίρεση των παραγόγων των ε, συναλλαγών ε, για την μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία έχουμε τοποθετηθεί ε, όσον αφορά αυτές τις εξαιρέσεις, προβλέπονται αυτές οι εξαιρέσεις και μπορούν να διατηρηθούν με την ε, συμπερίληψή τους. Αν λοιπόν διαφωνήσουμε, ε, απλά θα μπούμε σε μια άλλη είδους ρύθμιση από το παραθυράκι. Και ε, θέλω να σας πω, αυτό θα συνεπάγεται εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν κατά νου ότι η αξιολόγηση κινδύνων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κερδοσκοπία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πιστεύω ότι η συντονίστρια των σοσιαλιστών, η αξιότιμη κυρία συνάδελφος, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι αν συμφωνήσουμε ή όταν συμφωνούμε με το φόρο χρηματοψηφιστικών συναλλαγών, θα πρέπει να υπάρχουν και λογικές εξαιρέσεις. Το λέω αυτό με σαφήνεια. Και εδώ εντάσσονται και οι market makers. Ε, επίσης, ε, ορισμός του χρηματοψητικού Ινστιτούτου των συνταξιωτικών ταμείων ε, των εργαλείων της αγοράς χρήματος. Αυτά είναι πολύ λογικές εξαιρέσεις. Αν λοιπόν θέλουμε μια λογική τοποθέτηση θα πρέπει και οι συνάδελφοι από την άλλη πλευρά του Κοινοβουλίου να λαμβάνουν υπόψη στη δική μας γνώμη γιατί αλλιώς η ε, γνωμοδότηση που θα ε, προκύψει δεν θα έχει καμία αξία. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην Επιτροπή, στον ε, Διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας. Σας παρακαλώ όμως ε, να συντομεύσετε λιγάκι γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα στη μερίσια διάταξη και για τις 5 η ώρα ε, προβλέπεται ο κ. Μπαρνιέ. Θα σας ήμουν λοιπόν ευγνώμων αν μπορούσατε να μιλήσετε κατά το μέγιστο 3 λεπτά. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ, Πρόεδρε. Τώρα το θέμα είναι ποιο είδος μήνυμας πολιτικής θέλει να περάσει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ήδη έχουμε μιλήσει για το φορό χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όμως αν επιλέξετε το φόρο χαρτοσύμου μόνο, τότε πολλά δεν θα έπρεπε να μπουν στην έκθεση αυτή θα πρέπει πάντοτε να γνωρίζετε ότι όσο ε, περισσότερα από ή κάποιος, τόσο ψηλότερο θα είναι το κόστος για τους άλλους και τόσο πιο πολύπλοκο θα είναι να συλλεχθεί ο φόρος και τόσο περισσότερες ε, δυνατότητες θα υπάρχουν για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει να κάνει με τη φορολόγηση των συναλλαγών αυτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χρηματαγορές. Μιλάμε και για το σκιώδη τραπεζικό τομέα, όχι μόνο για τις τράπεζες ε, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε τα hedge fund, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους ΟΣΕΚΑ, αλλά Επίσης ε, σημαίνει και τους market makers, τους χονδρέμπορους χρηματιστηριακών συναλλαγών. Και θα ήθελα να αφαιρθώ εδώ σε τρία-τέσσερα πράγματα στα οποία αναφερθήκατε και εσείς. Καταρχήν το θέμα των χονδρέμπορων χρηματιστηριακών τίτλων και ε, το αποτέλεσμα συνεχών ε, συνεπειών. Όσοι το είπαν αυτοί πάντοτε θέτουν κατά μέρος τις διατάξεις του άρθρου 12, που λέει ότι αν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν ε, εξ ονόματο ενός άλλου ιδρύματος, μόνο το τελευταίος πρέπει να πληρώσει το φόρο, ενώ ε, θα πρέπει να μπουν εδώ και οι market makers. Το θέμα της εξοδευτικότητας είναι κάπως παράξενο για μένα, γιατί προέρχεται από αυτούς που ήταν κατά. Καταρχήν, ε, είμαστε κατά του φόρου γιατί είναι καλό για αυτούς που δεν συμμετέχουν και κακό για αυτούς που συμμετέχουν. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί που ανήκουν σε αυτούς που δεν συμμετέχουν και τώρα λένε είναι κακό για μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με την εξαίρεση ε, για ε, τις ε, δραστηριότητες που θα έπρεπε να υποστηριχθούν εδώ. Εδώ νομίζω η λογική δεν είναι απόλυτα σωστή γιατί πολλά από αυτά τα προϊόντα όπως τα τα ταμεία έχουν κάποιο προνομιούχα πρόσβαση στις κεφαλαγορές και λαμβάνουν κάποια εθνικά προνόμια όπως ε, μειωμένη επιβολή φορολογίας. Και έτσι λοιπόν αν υπάρχει ειδική μεταχείριση, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποια στομής, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και προνομία και μεταχείριση και στον τομέα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επίσης, ε, δεν ε, μπορούμε να μιλάμε για άσπρο ή μαύρο, δηλαδή για φόρο ή για εξαιρέσεις. Η κυρία για εξαιρεσεις η κυρια μετά αναφέρθηκε στις συμφωνίες ε, ΡΕΠΟ και ότι ίσως ε, θα έπρεπε να εξετάσουμε εκεί τη δυνατότητα μειωμένων ε, συντελεστών και όχι το συντελεστή που πρότεινε η Κομισιόν, θα το εξετάσουμε αυτό. Όμως κάτι τελευταίο, αν και ο κύριος Κλίντ φαίνεται να το αμφισβητεί, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα αποτέλεσμα κινήτρου στο κείμενο, γιατί τελικά ε, αυτοί που προβαίνουν σε συχνές συναλλαγές θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο. Είτε μιλάμε για εμπορευόμενους σε μεγάλη συχνότητα είτε για market makers. Ε, και κάποιοι που προβαίνουν σε μικρότερο αριθμό συναλλαγών θα πληρώσουν πολύ μικρότερο φόρο. Και επίση για τα συνδεξιωτικά ταμεία έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά προϊόντα. Κάποιοι ζητάνε τέλη εισόδου, εξόδου, διαχείριση επιδόσεων και αυτοί που προβαίνουν σε μεγαλύτερες τέτοιες συναλλαγές θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερο φόρο. Και αν τελικά επιλέξετε όλες αυτές τις εξερέξεις, τότε θα μειώσετε και το αποτέλεσμα του κινήτρου που υπάρχει στο κείμενο του φόρου με το πιστοτικών συναλλαγών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέγκμαν. Και να ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Ποδηματά. Thank you, Chair. Uh, it's impossible for me to deal uh, in each and Κοιτάξτε, είναι αδύνατο για μένα να τοποθετηθώ απέναντι σε όλες τις παρεμβάσεις. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδους ε, για τα σχόλιά τους. Κάτι άλλο το οποίο επιθυμώ να αναφέρω είναι το εξής. Περίπου αυτό που είπε και ο κύριος ε, Γκίγκολτ. Προς αυτή την κατεύθυνση τοποθετούμε. Δηλαδή το βρίσκω περίεργο το ότι οι αντίπαλοι του φόρου χρηματοψηφιστικών συναλλαγών σε παλαιότερες συζητήσεις ε, όταν μιλάγαμε για φόρο να επιβληθεί και σε 27 χώρες είχαν πει ότι ο φόρος ήταν πολύ άσχημα ε, σχεδιασμένος και αυτό θα οδηγούσε σε μεγάλης κλίμακας ε, φοροδιαφυγή. Και τώρα οι ίδιοι λένε ότι κάποια τμήματα αυτού του φόρου είναι τόσο καλά σχεδιασμένα που θα επιβάλλουν, θα συνεπάγονται αρνητικέ συνέπειες. Εγώ σας επαναλαμβάνω τη θέση μου. Είμαι ανοιχτή, απόλυτα ανοιχτή να συζητήσω ε, κυρίως ε, όταν πρόκειται για ε, βασισμένες και ουσιαστικές επιφυλάξεις. Αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο επουδενή δεν πρέπει να ανοίξει το παράθυρο προς διαφόρων μορφών εξαιρέσεις που θα υπονόμευαν όλο το οικοδόμημα που είχαμε σκεφτεί από την αρχή. Δηλαδή έναν ευρεία κλίμακα σε φόρο χρηματοψηφιακών συναλλαγών που θα καλύπτει όλες τις συναλλαγές, ε, όλες τις και όλες τι περιπτώσεις. Επίτρεψέ μου να σου πω πριν φύγεις όλε ότι αυτό κυρίως ήταν ο λόγος που απέτυχε ο φόρος αυτός στη Σουηδία. Δηλαδή περιορισμένη εμβέλεια και υψηλή φόρη. Άρα δηλαδή πρέπει να επωφεληθούμε από την εμπειρία που κάναμε στη Σουηδία. Όσον αφορά τώρα τις διάφορες εξαιρέσεις για τα ρέπος, ε, κύριε Μπέρκμαν, ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε και με το σχόλιο σας ότι η Κομισιόν ενδεχομένως να εξετάσει το ενδεχόμενο του χαμηλότερου φόρου του 0,01% σε ρέπος με μικρότερη διάρκεια. Πράγματι αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στα συνταξιωτικά ταμεία σε συναλλαγές μεταξύ ομάδων, intergroup ε, transactions και τέλος Όσον αφορά αυτό το περίφημο επιχείρημα της εξοδαφικότητας, εξοδαφικών ρυθμίσεων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η αρχή της μόνιμης κατοικίας επί της οποίας βασίζεται αυτή τη στιγμή η πρόταση, αυτή η αρχή της μόνιμης κατοικίας χρησιμοποιείται ευρέως σε θέματα φορολογικά και κατ' ουσίαν αυτή είναι και η αρχή που ισχύει και για τον φόρο προστέμενης αξίας. Με βάση λοιπόν ε, κανόνες του ΦΠΑ που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, όσοι χρησιμοποιούν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλουν το ΦΠΑ στη χώρα του αγοραστή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας Γερμανός αγοράσει online κάτι από την Amazon, η Amazon καλείται να καταβάλει το ΦΠΑ στις γερμανικές αρχές. Εδώ λοιπόν στο δικό μας το φόρο έχουμε τον ίδιο σχεδιασμό και εξ όσων γνωρίζω για το ΦΠΑ τουλάχιστον δεν προέκυψαν νομικές προσφυγές, αμφισβητήσεις. Επίσης, το θέμα του ε, φόρου χαρτοσύμου εφαρμόζεται από τις αγγλικές εταιρείες ανεξάρτητα από το που λαμβάνει η χώρα η συνδιαλλαγή και ανεξάρτητα με το αν μιλάμε για ε, Άγγλο υπήκο ή όχι. Και σας λέω ότι το 40% περίπου των φορολογικών εισόδων του Ηνωμένου Βασιλείου προκύπτει από αλλοδαπούς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα επιχειρήματα έχουν άμεση σχέση και ρυθμίζουν το θέμα της εξοδαφικότητας. Αυτός είναι ένας φόρος τον οποίο τον εγκρίνουν και σχεδιάζουν να τον εφαρμόσουν 11 κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι χωρίς να θέλω βεβαίως να εξαιρέσω τους ε, συναδέλφους ή τα κράτη-μέλη από τις δικές τους τις ε, συμβολές στο σχεδιασμό του φόρου εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στα κράτη-μέλη εκείνα που έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας αυτά να ε, κανονίσουν τις λεπτομέρειες του φόρου. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ. Ε, προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία με τους σκιώδης ηγητές, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να είναι ο θεσμός εκείνος που θα ανοίξει την πόρτα, που θα αντιμετωπίζεται απ' έξω ως ο θεσμός εκείνος ο οποίος ξεκίνησε την υπονόμευση, την οθή αν θέλετε, ε, του ε, φόρου χρηματοψηφιστικών συναλλαγών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αποδηματά. Στις 6 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και πάμε ταχύτατα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξης, σημείο υπαριθμών 5, στην περιφερειακή πολιτική. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε δει τις συμβιβαστικές τροπολογίες, δεν τις συζητήσαμε. Δεν γίνεται λοιπόν στις 6 Ιουνίου να ψηφίσουμε αν θέλουμε να τα κάνουμε τα πράγματα σοβαρά και να συμφωνήσουμε όπως είπε ο κύριος Φέρμπερ δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στις 6 αφού δεν έχουμε τίποτα από τα προτινόμενα μπροστά μας δεν μπορούμε έτσι να καταλήξουμε σε συνένεση λογική και δεξάλλου δεν επήγει το θέμα δώστε μας περισσότερο χρόνο ο Μιτεράν έτσι έλεγε πάντα πρέπει να δώσουμε χρόνο στο χρόνο Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ ο χρόνος, αλλά μου λέει η γραμματεία ότι οι συμβιβαστικές διανεμήθηκαν μεταξύ των σκιωδών, άρα οι πολιτικές ομάδες ήδη μπορούν να τις συζητήσουν. Ορίστε κύριε Ρόζες, Γκοζές. Κύριε Πρόεδρε, ως συντονιστής, δεν το επικαλούμε συχνά, αλλά εδώ γίνεται μία βλακώδης επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης. Αποφασίζουμε κάτι, τρεις μέρες αργότερα το αλλάζουμε γιατί δεν δόθηκε αρκετός χρόνος για τη διορία κατάθεση τροπολογιών. Αυτό δεν επιταχύνει τίποτα. Αφήσουμε χρόνο να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Αλλιώς είναι απλό το θέμα θα γίνουν όλα πρόχειρα αν δεν υπάρχει ο καταλληλότερος χρόνος, ο κατάλληλος χρόνος εμείς θα καταψηφίσουμε όποιο και να είναι το σχέδιο και η πρόταση. Και αυτό δεν βοηθάει κανέναν, κυρία Ποδηματά. Ναι, ένα σχολιάκι. Καταρχήν, οι συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν ήδη διανεμηθεί. Κυρία Λούλινγκ, ακούστε με ένα λεπτό. Εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα ζητούσα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως εισηγήτρια. Προγραμματίσαμε λοιπόν δύο νέες συναντήσεις με τους Κιώδης για να κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια συμβιβασμού. Τρίτον, και θέλω να το καταθέσω εδώ στους συναδέλφους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των κυρίων θέσεων Ζαμπόλ που έλαβε ήταν και η προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία για τον φόρο αυτόν πριν τις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι σημαντικό. Μα είναι σε ένα χρόνο. Ναι, αλλά είναι σημαντικό το κοινοβούλιο να παραμείνει συνεπές, τουλάχιστον το κοινοβούλιο με το στόχο αυτόν. Αυτή είναι η θέση μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρόεδρος. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε στις 10. 10 πώς σας φαίνεται. Θέλετε λίγες μέρες παραπάνω. 10 Ιουνίου είναι τη Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο. Ε, βέβαια η χειρότερη ώρα είναι αυτή. Αν δεν ψηφίσουμε στις 10 ε, θα αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Δεν προλάβουμε να ψηφίσουμε μέχρι τον Ιούλιο και αυτό είναι πρόβλημα και αρκετά μέλη επιθυμούν να το κλείσουν το θέμα πριν από το καλοκαίρι. Έχω λοιπόν την εντύπωση, λέω ότι καλύτερα ε, να τηρήσουμε τις προθεσμίες, να ψηφίσουμε στις 10. Αν δεν έχουμε ακόμα συμβαστικές προτάσεις κοντά σε αυτήν την Ρωμανία θα το ξαναδούμε. Έχουμε άλλη μια επιτροπή μέχρι τότε και μπορούν να έρθουν οι συντονιστές. Ο Ζαν Πολ ζήτησε και πάλι το λόγο. Πρόεδρας. Έτσι είναι, ίσως ε, να μας πιέζει για χρόνος, όμως καταλήξαμε σε αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα και σε επίπεδο κοινοβουλίου παίρνουμε αποφάσεις για να έχουμε ε, συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, να μην αποφασίζουμε πολύ γρήγορα και ταυτόχρονα τελικά οργανωνόμαστε με έναν τρόπο έτσι ώστε να μην μπορεί να τοποθετηθεί κανένα σκιώδης. Δεν έχουν χρόνο οι βουλευτές να συζητήσουν στην ομάδα το θέμα και ως συντονιστές πρέπει να συμφωνούν και οι υπόλοιποι συναδελφοί αν ε, εργάζονται κάποιοι σκιώδεις ε, για το φακέλο πολύ ωραίο όμως ε, ε, σε κάποιες συνεδριάσεις ε, εμφανίζονται κάποιοι συνάδελφοι να λένε ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την Επιτροπή πάντοτε θέλαμε τη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση και τώρα δυστυχώς τους βλέπουμε να μην έχουν και χρόνο οι σκιώδεις. Σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογέ είναι σε ένα χρόνο. Εγώ είμαι βουλευτής μέχρι την τελευταία ημέρα της θητής και μέχρι τότε θα δουλέψω. Ευχαριστούμε κύριε Κουσές. Σβέν, πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το θέμα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα ως προς το χρόνο. Δηλαδή, αν κάποια μεγάλη ομάδα ζητούσε περισσότερο χρόνο, δεν είχαμε ποτέ κόλλημα στο να παράσχουμε το χρόνο αυτό. Θα πρέπει οι σκιώδεις συνήθως να μπορούν να συμφωνούν σε ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα και λυπάμαι που στο Συμβούλιο δεν βλέπω να υπάρχει κίνδυνος να το ολοκληρώσουν αυτό πριν το καλοκαίρι. Δυστυχώς θα ήθελα ένα γρήγορο αποτέλεσμα, αλλά δεν βλέπω και μεγάλη πολιτική αξία. Επομένω, συμφωνώ με πολλά πώ υπόθηκαν να συρεμήσουμε. Έχουμε πάρα πολλέ ευθύνε σε αυτή την εντολή, σε αυτή τη θητεία, με συγχωρείτε, και τα περισσότερα που κάνουμε σε αυτό το κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρουν κανέναν από του πολίτε. Και δεν καταλαβαίνω εδώ ότι θα έπρεπε να λειτουργήσουμε διαφορετικά επειδή έχουμε τις ευρωεκλογέ. Πρέπει να νομοθετήσουμε και χρειαζόμαστε ένα πνεύμα συνεργασίας. Ας μην το καταστρέψουμε λοιπόν αυτό. Εγώ εμπιστεύομαι ότι θα μπορούν να βρουν μια καλή λύση σκιώδης και εισηγήτρια για όλους. Και ας τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν είναι πρέπουσα να γίνεται εδώ. Και βλέπουμε κάποια ανησυχία ότι κινούμαστε σε ένα μόντο εκλογικό. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε την ικανότητά μας να υλοποιήσουμε τα καθήκοντά μας. Ευχαριστούμε κύριε Γκίκολτ. κύριε Σλάνγκερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πού καταλήγουμε όταν αναγκαζόμαστε να λάβουμε πολλές αποφάσεις στο Στρασβούργο. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίζαμε από τις 9 παρτέτο μέχρι τις 10.30 για την έκθεση Χόκμαν. Και αυτό πραγματικά ήταν υπερβολική απέτηση. Εμείς και την προηγούμενη θητεία και αυτήν ε, είπαμε ότι δεν γίνεται να γίνονται όλα αυτά στο Στρασβούργο. Η 10 του μηνός είναι Δευτέρα στο Στρασβούργο και ε, ο πρώην πρόεδρος ε, αρνείται να το κάνει αυτό και τώρα τα εγκρίνει όλα. Όποιος λοιπόν θέλει να έχει κάποια έγκριση ως πρόεδρος για το Στρασβούργο την παίρνει. Αυτό λοιπόν είναι αντιφατικό και δεν είναι σωστό. Δεύτερον, η έκθεση Μακάρτη ε, αναβλήθηκε γιατί δεν είχαν κατατεθεί οι σημαντικές προτάσεις και, και αν είχαν κατατεθεί δεν συζητήθηκαν. Γιατί δεν κάνουμε και εδώ το ίδιο. Η 17η, 18η είναι μια χαρά, και εκεί μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς να υπάρξει ουσιαστική χρονική καθαστέρηση. Πρόεδρο, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λάγκη να δώσω το λόγο στην Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Κοιτάξτε, εγώ γενικά ε, το να αναβάλουμε ε, είμαι ανοιχτή. Όποτε είναι απαραίτητο και σημαντικό κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε βέβαια να το αποφασίσουμε τώρα. δεν μπορούμε τώρα να αποφασίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω η συγγήτρια και οι σκιώδεις ε, να συμφωνήσουν, αλλιώς θα πρέπει να ψηφίσουμε για την ε, αναβολή. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος ε, για να λυθεί το θέμα. Ελπίζω όμως ε, πριν ψηφίσουμε αύριο να μου καταθέσετε, να μου πείτε ότι συμφωνήσετε γιατί αλλιώς τι να κάνω κι εγώ ε, θα πω να αναβληθεί η ψηφοφορία και όλα αυτά τα χειριζόμαστε δημοκρατικά στην Επιτροπή μας. Είναι βέβαια πρόβλημα ότι ε, κάποια μέλη ομάδων δεν μπαίνουν έγκαιρα προτάσεις. Δεν πρόκειται μόνο την έκθεση, πρόκειται γενικότερα για πάρα πολλές εκθέσεις. Η Κομισιόν, ο Επίτροπος μάλλον, έχει έρθει για να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί του. Ας το κλείσουμε το θέμα. Βρέστε τα κάπως και πέστε μου αύριο που καταλήξατε. Και τώρα ε, γίνομαι, ξαναπαίρνω πάλι ε, την θέση της Πρόεδρου. Ε, το θέμα μου θα συζητηθεί αύριο. Ε, ψηφιστεί αύριο. Θα σας στείλω σε γραπτή μορφή τα σχόλιά μου και ελπίζω αυτό να φτάνει. Right, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαρνιέ θα πρέπει να φύγει ακριβώς 6 και 4 γιατί πρέπει να μεταβεί στο Άμστερνταμ. Επομένως ε, δεν θα χρονοτρεβήσουμε τώρα σε εισαγωγικά σχόλια. Είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος επίτροπος στην Επιτροπή μας. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα κατευθείαν να σας δώσουμε το λόγο και κατόπιν να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ Μισελ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας και τα πρώτα μου λόγια Σαρού θα είναι για να σας ευχαριστήσω για την κατανόησή σας. Και εγώ σας ζήτησα να μεταφέρετε χρονικά αυτή την ε, συνάντηση κάποιες μέρες, ε, γιατί εδώ και τέσσερις εβδομάδες ε, είχε προγραμματιστεί ένα χειρουργείο. Έτσι λοιπόν πριν 15 μέρες δεν ήμουν σε θέση να εμφανιστώ στην Επιτροπή σας. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, βρισκόμαστε σε μια βασική περίοδο της κοινή μας δράσης Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Ένα έτος μετά, με πριν το τέλος της εκλογικής ε, σίγουρα Πρέπει να γίνει κάποιο, απολογισμός, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερη σημασία στις προτεραιότητες που θέτουμε, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν κάποια απαραίτητα κείμενα τους επόμενους ε, μήνε. Ε, πολλά κάναμε τα τελευταία τρία έτη από κοινού και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που συμβάλατε σε αυτή την πρόοδο. Και φυσικά να πω ότι πολλά απομένουν να γίνουν, είναι σημαντικές οι προσδοκίες, είναι μεγάλες οι προσδοκίες και μαζί με την ε, κυρία Σάρον Μπόουλ στο τύπο συμβουλίου Κοφίν στο Δουβλίνο ε, το διαπιστώσαμε αυτό και στις τελευταίες συνεδρίες της G20. Επίσης έχουμε επικεντρωθεί σε τρεις φακέλους που δεν είναι οι μόνοι. Η Τραπεζική Ένωση για την ταχεία ε, θέσπιση του συστήματος εξυγένσης των ε, τραπεζών, ε, την ολοκλήρωση του έργου του ρυθμιστικού μας και επίσης τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε κάποιες ρυθμίσεις ε, που ε, θα έχουν να κάνουν ε, όχι τόσο με την επανόρθωση των αποτελεσμάτων της κρίσης αλλά με την πρόληψη και μια νομοθεσία που θα, είναι, θα δώσει δυναμισμό στην ανάπτυξη. Λοιπόν, για την ε, Τραπεζική Ένωση κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη αρχικά ή μάλιστα και ουτοπική. Τώρα γίνεται πραγματικότητα με δύο κυρίους πυλώνες, την εποπτεία και ε, την εξυγίανση των τραπεζών και την εγγύηση των καταθέσεων. Χάρη στην ε, δουλειά του συγητή σας, του κ. Γκίκουλτ, είναι σε καλό δρόμο η εποπτεία. Συζητήσαμε το θέμα ε, της στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο και ελπίζουμε να υλοποιήσουμε το έργο μας και σε καθεστώς δημοκρατικών εγγύσεων. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα της εξυγίανσης. Η κρίση της Κύπρου μας επιβεβαίωσε ότι δεν είναι θεωρητικές αυτές οι ανησυχίε και θέλω να ευχαριστήσω και τον Γκούναρ Νότμαρκ ε, που είναι ο σκιώδης ε, εισηγητής για το θέμα αυτό για την οδηγία της εξηγένσης των τραπεζών. Και νομίζω ότι οι τριμερείς διάλογοι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε κάποια θέματα κλειδιά που συζητήθηκαν και από τους υπουργού πριν λίγες ημέρες, τη χρηματοδότηση της εξηγένσης, την διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάσωση με ίδια μέσα, με τον bail-in. Και τη συμμετοχή των πιστωτών και την ημερομηνία εφαρμογής. Σε λίγες μέρες, τον Ιούνιο, θα παρουσιάσουμε μία πρόταση ενίως μηχανισμού για την εξυγένση των τραπεζών στην Ευρωζώνη και θα υπάρχει ένα κοινό ταμείο εξυγένσης που θα προχρηματοδοτείται από τις τράπεζες και την πρόταση μιας αρχής εξυγίανσης που θα θέτει σε εφαρμογή τους κανόνες της οδηγίας εξυγίανσης των τραπεζών της Ευρωζώνης. Ελπίζω ότι αυτός ο πλήρης μηχανισμός θα μπορέσει να λειτουργήσει παράλληλα με την εποπτεία το 2014. Αλλά θα έχουμε την πλήρη λειτουργία του μηχανισμού σίγουρα το 2015 πέρα από την Τραπεζική Ένωση. Ε, το έργο της ρύθμισης ε, είτε για να διορθωθούν τα λάθη είτε για να προληφθούν κάποιες καταστάσεις ε, συνεχίζεται. Έχουμε κάνει καλή πρόοδο από κοινού και ευχαριστώ τον Βέρνερ Λάγκεν για την ε, έγκριση της σχετικής έκθεσης για τα παράγω και τον Ότ Μαρκάρας και για το πακέτο της Οδηγίας Κεφαλαϊκών Απαιτήσεων 4. Έχουμε επίσης συζητήσεις για τρεις πολύ σημαντικούς φακέλους με τον Μάρκο Φέρμπερ για το φάκελο MIFID, επί του οποίου θέλουμε να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο των συντομότερο δυνατών και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα ακόμη μεγαλύτερη αφού παρόμοιοι κανόνες ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επουσία ενός Leven Blankfield field είναι κάτι που θέτει δυσκολίες σε όλες τις επιχειρήσεις ε, και εδώ αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο δεύτερος φάκελος είναι κατά κατακρίσει στην αγορά. Χαίρομαι για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για ένα φιλόδοξο κανονισμό που θα ενισχύσει το νομοθετικό μας πλαίσιο. Και τέλος ε, θα πρέπει με τον Μπόρκαν Μπάλ στο συντομότερο δυνατό να συνεχίσουμε τον τριμερό διάλογο για το Omnibus 2 ε, καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί οι πρόσθετες μελέτες για τα ασφαλιστικά προϊόντα με τις μικροπρόθεσμες εγγύσεις. Τώρα, αναφέροντα ε, εντάχει αυτού ε, του τρει φακέλου, δεν υποτιμώ τη σημασία άλλων φακέλων που είναι επιτάπητος, ε, του ΟΣΕΚΑ 5, ο ε, είναι η στην διαμεσολάβηση ασφαλιστικών προϊόντων, Βέργεν Λάγκεν και τα ΠΡΙΠΣ με την περιβάλληση Μπέρε ή το CSD με την Κέσ Πίτνερ. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν μόλις παρουσίασε μια οδηγία πολύ σημαντική για μένα, για την επιμήκυνση της έκθεσης του Κλούτε το 2011 που έδωσε ε, πρόσβαση σε όλους τους Ευρωπαίους σε ένα βασικό λογαριασμό στην τράπεζα για να βελτιωθεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των τραπεζικών εξόδων και να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Ξέρω ότι ε, υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά, πολλοί φακελοί ανοιχτοί και υπάρχει πολύ μεγάλο άχθος εργασίας. Αυτός όμως είναι ένας λόγος να σταματήσουμε, όπως ε, θα ήθελαν ε, κάποιοι φορείς των χρηματοπιστωτικών αγορών, δεν το πιστεύω. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε νέες δυσλειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σκέφτομαι ιδίω την υπόθεση που αποκαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο για τους ε, δείκτες αναφοράς. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τις συνέπειες ε, της υπερβολικής ρύθμισης που δεν θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύσει ε, στα συγκοινωνούντα δοχεία το παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Αυτά τα δύο θέματα και καθώς για το θέμα της ελευθερίας οδηγίας για τις ε, υπηρεσίες πληρωμών ε, θα σας ε, πρότεινα να το δούμε πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους συστημικούς κινδύνους που δεν, θα, δεν θα λαμβάνονταν υπόψη από τα μέτρα ρύθμισης και μιλάμε για την διαρθρωτική ρύθμιση των τραπεζών. Πρόταση που θα παρουσιάσω αμέσω μετά το καλοκαιρινό θέρος κατόπιν της έκθεσης Λικάνεν. Θα ξεκινήσω μια συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Καρτή για την έκθεση πρωτοβουλίας που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε μια σχετική φιλοδοξία για το θέμα αυτό. Επίση, για το φθινόπωρο θα προτείνω αναθεώρηση τη οδηγία για τα συνταξιδετικά ταμεία για να προστατεύσουμε καλύτερα του ασφαλισμένου και να βελτιώσουμε τη λειτουργία τη ενία αγορά. Όπω είπα πρόσφατα στο Άμστερνταμ, αυτή η αναθεώρηση καταρχήν ε, θα θίξει ε, το θέμα τη διαφάνεια, τη διαχείριση και του reporting τη σημερινή οδηγία. και σε δεύτερο χρόνο θα ασχοληθούμε με τι απαιτήσει προληπτική εποπτείας γιατί ε, ο πρόεδρος του ΙΟΠΑ με ενημέρωσε για τις δικές του ανάγκες, ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αξιολογηθούν καλύτερα οι ποσοτικέ εγγυήσει για τα στεξιωτικά ταμεία. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα αυτό και εγώ δεν θέλω να διακυβευθεί η κατάσταση των συνταξιδοτικών ταμείων μακροπρόθεσμα. Και για να κλείσω, ένα, κάτι τελευταίο σχετικά με το θέμα της αναγκαιότητας. Φέτος είναι ένα έτος κλειδί για να ολοκληρώσουμε αυτά τα κείμενα. Δηλαδή μίλησα για κάποια νομοθεσία προληπτική, διορθωτική ε, και πρέπει να περάσουμε αυτή την διορθωτική νομοθεσία σε μια πιο προληπτική νομοθεσία, να εκδομήσουμε την Τραπεζική Ένωση και να θέσουμε σε εφαρμογή τις αποφάσεις της αυτά είναι σημαντικά, αλλά έχουμε τώρα την ευκαιρία να ρυθμίσουμε και το παραγωγικό κεφάλαιο, όχι μόνο το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και αυτό θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα προϊόντα. Γνωρίζετε την πράσινη βίβλο που δημοσιεύσαμε πριν ε, λίγες εβδομάδες ε, για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επίσης ε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα δημοσιονομικά θεστώτα, πρέπει ε, να ρυθμίσουμε, να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση από τη, την τραπεζική ή τη μη τραπεζική, να υπάρχει προώθηση της καινοτομία, όλες αυτές τις ιδέες λοιπόν τις έχουμε θέσει στη συζήτηση και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Και κάτι τελευταίο, συμπερασματικά, κατόπιν των συμπερισμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ε, στην ε, περίπτωση του reporting, της υποβολής εκθέσεων, θα έχουμε ε, καλύτερες συνθήκες διαφάνειας για τους φόρους που έχουν καταβληθεί. Αυτά έχουν εισαχθεί για τις τράπεζες στο πλαίσιο της CDR4, της Οδηγίας Κεφαλαιών Κοπετήσεων 4. της οδηγιας κεφαλαιων πεπισεων 4 επομενως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και πώς, ποιοι είναι οι φόροι που καταλάβουν και εξορρυκτικές βιομηχανίες ε, ή οι βιομηχανίες που ασχολούνται με τη δασοκομεία και στο θέμα της ε, φορολογίας όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να δηλώσουν διαφανώς τι καταβάλουν, ποια ποσά και σε ποιου. Και αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε, στο χρόνο που είχα πριν ε, να σας ακούσω και να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. ευχαριστώ και για την προσοχή σας, αλλά και για τη συνεργασία. Σα Σας κατευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Με μεγάλη χαρά άκουσα αυτά που είπατε για τις αναφορές οι μελέτες χώρα με χώρα. Δεν έχουμε ακόμη οδηγίες για τη διαφάνεια ως προς αυτά και θα ήταν ο πιο σύντομος τρόπος να εφαρμοστούν οι ιδέες αυτές γιατί και το Συμβούλιο είχε πει ότι για τις μη δημοσιονομικές αποκαλύψεις πρέπει να ό,τι προταθεί να γίνει με τρόπο που να συμφωνεί με την οδηγία για τη διαφάνεια των λογιστικών. Τώρα, θα χρειαστεί να μειώσουμε τους χρόνους για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Τέσσερα λεπτά για την ερωταπάντηση. Και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να θέσει ερώτηση πάνω από δύο λεπτά. Αλλιώς δεν θα ακούσει απάντηση. Και οι πρώτοι και οι τελευταίοι θα σεβαστούν αυτό τον κανόνα γιατί πρέπει κάποτε να φύγει και ο Επίτροπος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Μαριάννα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας και για όσες πληροφορίες μας δώσατε. Θα επισέλθω αμέσως στην ουσία. Μας ανακοινώνουν συχνά ότι θα υπάρξει μία single resolution authority λένε. Μήπως θα μπορούσατε να μας αποκαλύψετε τουλάχιστον μέχρι κάποιον βαθμό πώς η ευρωπαϊκή αυτή αρχή θα είναι κάτι παραπάνω από έναν απλό συντονισμό εθνικών αναλόγων αρχών. Τι παραπάνω θα κάνει δηλαδή, ώστε πράγματι να κρατάει τα ηνία των εξελίξεων. Ελπίζω να μας πείτε με τι εργαλεία, με τι μέσα θα το πετύχετε και αν θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο financial backstop. Μήπως λοιπόν είστε περιορισμένοι, σας περιορίζουν οι συνθήκες, μήπως αυτά που θα θέλατε να γίνουν δεν θα μπορέσετε να τα εφαρμόσετε κατά τη θητεία τουλάχιστον αυτή της Κομισιόν. Και η Κομισιόν είναι ή όχι σε θέση να κινήσει τα πράγματα ώστε να γίνει κάποια πρόοδος εφόλων αυτών. Κοιτάξτε, αν μου το επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε να επανέλθω σε κάτι που είπατε εσείς προηγουμένως για τη διαφάνεια που την υποστηρίζω και εγώ. Οι μεγάλες εταιρείες και το τι πληρώνουν φορολογικά Επ' αυτού δεν έχω καμιά συγκεκριμένη ιδεολογία για το πότε ακριβώς πρέπει να εφαρμοστεί η ρήτρα αυτή. Είμαι υπέρ, θα ήθελα να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα και με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια. Δεν έχω λοιπόν προκαταλήψεις και προκαθορισμένες ιδέες. Με οποιοδήποτε μέσο, είτε δηλαδή με το κείμενο για την οδηγία της διαφάνειας, είτε και για το θέμα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και της περιβαλλοντολογικής, αλλά όσο το δυνατόν συντομότερα και όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Αυτό. Και τώρα επανέρχομαι στο ερώτημα της Μαριάν Τίσεν. Θέλω να απαντάω συγκεκριμένα, αλλά ταυτόχρονα να βλέπω και τι άλλο συζητούμε στην Κομισιόν. Εγώ συνεργάζομαι πολύ με τον πρόεδρο Μπαρόσο και με τον συνάδελφό μου Όλη Ρεν καθώς και με τον συνάδελφο Αλμούνια που ασχολούνται από διαφορετικές οπτικές ο καθένας με τις τράπεζες. Θα πρόκειται για μια ενιαία αρχή που θα εργάζεται παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή όπως ζητήσατε κι εσείς. Και θα προβλέψω διατάξεις βάσει των οποίων η ενία αυτή αρχή θα αφορά και τις χώρες που δεν έχουν ακόμη μπει στην Ευρωζώνη αλλά που θα ήθελαν λογικά να συμμετέχουν στην εποπτεία θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από μια, έναν απλό συντονισμό γιατί τα όρια του συντονισμού τα έχουμε δει. Θυμάμαι όπως και εσύ σίγουρα την περίπτωση της Δέξια όπου τρεις χώρες χρειάστηκε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να αυτοσχεδιάσουν. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Θα πρόκειται λοιπόν για μια ολοκληρωμένη πραγματική αρχή με πραγματική δυνατότητα λήψης αποφάσεων με δημοκρατικό βέβαια έλεγχο και γιατί μιλάω για κοινό μηχανισμό για αυτή την αρχή γιατί η Κομισιόν έχει δίκιο που προτείνει την ευρωπαϊκότερη δυνατή το ευρωπαϊκότερο δυνατό επίπεδο για την εποπτεία. Αυτή η ολοκληρωμένη λοιπόν η ενιαία αρχή, κυρία Μαριάν Τίσεν, θα βασίζεται στην εργαλειοθήκη του ψηφίσματος Γκούναρ Χόκμαρκ που θα το εφαρμόσουμε πλήρως. Και ξέρω ότι συζητιέται και η έκθεση για τις εγγυήσεις των πληρωμών έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε πλήρως όλα αυτά τα εργαλεία για τις εγγυημένες καταθέσεις, για τις εγγυήσεις των καταθέσεων. Όλα αυτά πρέπει να έχουν κάποιο κοινό μηχανισμό που να συνδυάζεται με το μηχανισμό σταθερότητας. Ευχαριστούμε. Και τώρα... Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η ερώτησή μου Ακολουθεί την ερώτηση της κυρίας Τίσαν. Στο το Κοινοβούλιο όταν εκπώνησε τη θέση του για την τραπεζική εξυγίανση έδωσε προτίμηση στην ιεραρχία του Μπέιλιν στους καταθέτες ακόμη σε αυτούς που είναι άνω των 100.000 ευρώ. Πάνω από τα 100.000 ευρώ η αρχή εξυγίανσης ε, ε, μήπως ε, θα μπορούσε να μοιάζει με κάτι που έχουμε στις ΗΠΑ με το ρόλο του FDIC για να διασωθούν οι καταθέσεις, γιατί εγώ νομίζω το Μπελίν δεν είναι το κατάλληλο μέσο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις καταθέσεις και εγώ νομίζω ότι η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών ε, εξαρτάται πάρα πολύ από το να κατανοήσουν τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση αυτή, να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Να ξαναπώ και να επιβεβαιώσω υπό το φως των λαθών των προβλημάτων ε, που συναντήσαμε στη διαχείριση της κυπριακής κρίσης, ότι σε όλες τις περιπτώσεις παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ θα πρέπει πάντοτε να εγγυώνται. Αυτή είναι μια διασφάλιση που την αφήλουμε στους αποτεμιευτές σε κάθε περίσταση. Γιατί στο κείμενό μας προβλέψαμε από την αρχή γιατί το κείμενο για την εξυγίανση και τη διαχείριση της τραπεζικής κρίσης σας το έχω προτείνει εδώ και ένα χρόνο. Και τότε δεν άκουσα και πάρα πολλά σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί ο στόχος ήταν να βρούμε από κοινού τα μέσα ανακοινώνοντα σε όλους από την αρχή του κανόνε του παιχνιδιού ότι οι τράπεζες πληρώνουν για τις τράπεζες και όχι οι φορολογούμενοι, όπως είδαμε να γίνονται τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπου οι φορολογούμενοι, χωρίς να τους ζητάμε και τη γνώμη του, κλήθηκαν να πληρώσουν για τη διάσωση των τραπεζών. Έτσι λοιπόν ε, το θέμα των καταθετών άνω των 100.000 ευρώ και τη δυνατότητα που θα υπήρχε να κληθούν ε, να καλύψουν ένα μέρος της απώλειας ε, μπήκε στη συζήτηση και γι' αυτό στη συνάντηση που είχαμε με τους υπουργού πριν λίγες ημέρες υποστηρίξαμε να σκεφτούμε το εξής μία πιθανότητα να τους δώσουμε μία προνομιούχο σειρά ε, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις απολιές τους. Δηλαδή μιλήσαμε για τους ε, μετόχους, ε, για τους πιστωτές, τον τάδε και το δίνα και στο τέλος να μπουν οι καταθέτες που έχουν καταθέσει άνω των 100.000 ευρώ. Αν τελικά συμφωνήσουν οι νομοθέτες, δηλαδή εσείς και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό, για το σημείο αυτό, νομίζω ε, θα μπορούσαμε να τους βάλουμε στο τελευταία σειρά ε, της ιεραρχίας. Δηλαδή να είναι οι τελευταίοι που θα κληθούν ε, οι καταθέτες. Και όπως σας είπα, για τους μικρούς ε, καταθέτες δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί υπάρχει εγγύηση. Όμως θα μας πέτρεπε οι καταθέσεις άνω των 100.000 να διατηρηθούν και αυτή η προτίμηση θα μας επέτρεπε να έρθουν να συνεισφέρουν οι καταθέτες αφού θα έχουν συνεισφέρει στη διάθεση της τράπεζας όλοι οι προηγούμενοι. Έτσι λοιπόν εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε τελικά το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει με τέτοια πρόταση προτίμησης. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εσείς ε, Δικαίως αναφέρεστε σε ένα βαρύ πρόγραμμα εργασίας ε, και εμείς ε, προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί όλα τα αριθμιστικά μέτρα που εμείς εγκρίναμε από κοινού έχουν νόημα. Όλα έχουν νόημα και γνωρίζουμε γιατί αποφασίσαμε τόσο αποφασίσαμε. Όμως ε, το σωρευτικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιγότερο θετικό γιατί δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε αν προσπαθήσετε να δείτε ποιο θα είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα όλων των μέτρων που εμείς ε, αποφασίσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, αλλά μας το υποσχεθήκατε πριν ένα χρόνο ότι θα το πράξετε. Και μάλιστα είδαμε ότι πολλά από τα μέτρα σε πολλά από τα μέτρα τα κράτη-μέλη ήδη ε, λαμβάνουν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Στη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, έχουμε κάποια μέτρα που εφαρμόζονται στο τραπεζικό σύστημα, το ίδιο ισχύει και στο Ενωμένο Βασίλειο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει τα δικά της νομοθετικά, τις δικές της νομοθετικές ε, προτάσεις, ε, όμως ε, το ότι υπάρχει αυτή η διάκριση μας εμποδίζει στο να φτάσουμε σε κάτι ομοιόμορφο. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό στο μέλλον. Η ερώτηση του κυρίου Κλίντ είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί ακριβώ αναφέρεται στο επίκεντρο στο οποίο αναφέρθηκα και εγώ προηγουμένω ότι μπορώ το να έχουμε κάποια ε, ρύθμιση διορθωτική ίσως και κατασταλτική. Ε, δηλαδή αυτό πρέπει να το κάνουμε έχοντας κατά νου το τι έχει συμβεί και επίσης πρέπει να έχουμε και προληπτική ρύθμιση για να είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε θα θέτουν ισχυρά θεμέλια στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, χωρίς ε, ε, να εμποδίσουν την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Γι' Ε, θέλουμε κάποια μέτρα αξιολόγησης ε, της κάθε πρότασης. Για κάθε πρόταση υπάρχει μελέτη αντικτύπου, μελέτη αξιολόγησης και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Έχω κάποια παραδείγματα κατά νου και συχνά τα έχουμε συζητήσει και από κοινού για την οδηγία κεφαλαϊκών απαιτήσεων 4 ήμουν ένας από τους πρώτους, θυμάμαι ε, και πώς απευθύνθηκα στον τύπο για να ε, προειδοποιήσω για τα πρώτα προβλήματα ρευστότητα ε, και ο Μπερνάν είχε την ίδια θέση με μένα, το ίδιο είπε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τελικά τα... Ε, υπήρξε κάποια διόρθωση από την Επιτροπή της Βασιλείας. Επίσης, άλλο παράδειγμα για τις μακροπρόθεσμες εγγύσεις και άλλο παράδειγμα για τα συνταξιδοτικά ταμεία, όπου η ΟΠΑ μας λέει ότι χρειάζεται παραπάνω μήνες για να κάνει αυτές τις μελέτες αντικτύπου. Επίσης, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα αποτελέσματα που θα έχουν όλοι αυτοί οι νόμοι, ο ένας σε σχέση με τον άλλο. Και Γι' αυτό ε, θα έχουμε και αυτή τη δημόσια διαβούλευση μέσω της πράσινης βίβλου, γιατί θέλουμε να έχουμε μία συνολική εικόνα όλων των φορέων. Και επίση, ε, με το Wolfgang Klintz εργαζόμαστε για μια ε, πιο καθολική μελέτη που θα την κάνουμε όταν έχουμε μπει πραγματικά στις λεπτομέρειες για καθένα από τα νομοθετήματα αυτά. Όμως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τις συνέπειες αυτού του νόμου και για τα σωρευτικά αποτελέσματα γιατί δεν θα υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση της οικονομίας. Και ποιος θα χρηματοδοτήσει την οικονομία γιατί δεν είναι πλέον τα κράτη αυτά που μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι ο τόσο μικρό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ταπεινό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα το κάνει, αλλά είναι οι τράπεζε, τα συνταξιδοτικά ταμεία και οι αγορέ χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Και Αυτά τα θέματα τα έχω θέσει στην πράσινη βίβλο. Επίσης, ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε μία τρίτη ε, αξιολόγηση, να δούμε τι θα συμβεί και ε, με τους συνεταίρους μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και με άλλους ε, φορείς χρηματοπιστωτικούς ε, που δραστηριοποιούνται εδώ στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν θέλουμε να έχουμε ίσους κανόνες για όλους και γι' αυτό ε, συζητάμε με τους Αμερικανούς τόσο πολύ γιατί το 80% των συναλλαγών είναι υπερατλαντικές, διατλαντικές με συγχωρείτε. Thank you. Thank you, Commissioner. I'd like to... Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θέλω να φερθώ σε ένα από τα τελευταία θέματα που αναφερθήκατε, δηλαδή στην διατλαντική μορφή των διαπραγματεύσεων. Να σας ρωτήσω κατά πόσο μπορείτε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς γίνεται με την νομοθεσία ΕΜΠΗΡ σχετικά με τα παράγωγα. Ε, οι εφημερίδες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε διέξοδο ε, και προφανώς υπάρχει και άσκηση ποιησης και από τις δύο πλευρές, από ομάδες ποιησης. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας ενημερώσετε, θα ήμουν ευγνώμων. Και επίσης, εφόσον πρόκειται για Παγκόσμια Συμφωνία των G20, ε, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων των G20 απέναντι σε άλλες περιοχές, κυρίως απέναντι στην Ασία. Ε, τι ακριβώς γίνεται με την αναγνώριση τρίτων χωρών στις ασιατικές αγορές. Και επίσης ε, Μήπως μπορείτε να μας πείτε λιγάκι πού ακριβώς πιστεύετε ότι θα έχουμε φτάσει ε, μέχρι το τέλος της θητείας μας σχετικά με τα μεγάλα θέματα των αγορών. Ε, κυρίως εκεί που ε, από πέρυσι υπάρχει θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω κάποιος είπε έχει σχεδόν ξεχαστεί το περιεχόμενο γιατί έχει πια περάσει πολύ καιρό. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει αν θα ολοκληρωθούν τα θέματα μέχρι το τέλος της θητείας μας μας επίσης για τις καταχρήσεις αγοράς, για το CSDR ε, και επίσης και σχετικά με τις ασφάλειες, την ασφάλεια γενικότερα που τίθεται επιτάπητος. Αυτά είναι πολλές ερωτήσεις μαζί, θα απαντήσω τηλεγραφικά. Σας είπα ότι για το Μιφίντι ασχολούμαι και εγώ. Στο τελευταίο ΕΚΟΦΗΝ στις Βρυξέλλες πριν από μερικές μέρες η Ιρλανδική Προεδρία επέμεινε στα δύο εκρεμή θέματα και τα γνωρίζει ο κύριος Φάρμπερ, δηλαδή η διαφάνεια και η πρόσβαση. Και για μένα είναι και τα δύο σημαντικά, όχι μόνο το δεύτερο, για να είμαι ειλικρινής. Ελπίζω λοιπόν με την Ιρλανδική Προεδρία και την επόμενη τη Λιθουανική να επιδειχθεί απαιτούμενη πολιτική θέληση για να λυθούν και αυτά τα δύο πριν τη λήξη του έτους. Επίσης, για τις καταχρήσεις που μπορεί να σημειώνονται στις αγορές και αυτό έχει αρχίσει να συζητιέται και μπορεί να λυθεί και αυτό σύντομα για τα παράγωγα προϊόντα εξάλλου ιδιαίτερα. Η Διατλαντική Συμφωνία είναι μεν σημαντική αλλά δεν αρκεί. Γιατί εδώ μιλάμε για δοσοληψίες που αφορούν 600 εκατομμύρια, 600 χιλιάδες εκατομμύρια λέει ο ομιλητής, δηλαδή 600 δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. εκατομμύρια. Δεν είναι κάτι ασήμαντο λοιπόν. Γι' αυτό συζητώ και με τους αντίστοιχους στην Κίνα και αλλού για να το λύσουμε. Σας είπα λοιπόν ότι κάνουμε διεθνείς συνεννοήσεις συμμετέχουμε και στην ομάδα συντονισμού και επιτήρηση των παραγόγων προϊόντων που γίνεται, συναντιέται συχνά στις Βρυξέλλες. Έχω πάει πολλές φορές, επιτηρεί, εποπτεύει τον κόσμο ολόκληρο και έχει αναφερθεί στη δυσκολία που μπορεί να αντιπροσωπεύουν οι έλεγχοι αυτών των παραγωγών. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί εκεί πρόοδος, πολύ αργό μάλλον γιατί οι Αμερικανικές αρχές, η CFTC, δεν δέχεται να επεκταθεί και στις διαμεθοριακές δοσοληψίες η εποπτεία και ο έλεγχος. Όσο για την Κίνα, τις επόμενες μέρες προβλέπω συνεργασία και μαζί με τους Υπουργούς Οικονομικών της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Ιαπωνίας, της Ρωσίας, της Βραζιλίας και της Νότιας Αφρικής έχω απευθύνει στον ε, νέο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τις ανησυχίες μας, σε επιστολή του έχω απευθύνει. Καλά, ο Σβέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, ένα από τα κυριότερα στοιχεία της νομοθεσίας για τις κοιόδεις τραπεζικές δοσοληψίες Υποτίθεται ότι θα είχε υποβληθεί νωρίτερα, αλλά δυστυχώς έχει αλλάξει η ημερομηνία δημοσίευσης. Το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει δηλώσει ότι θέλει να σταματήσει πια η πρακτική του CNAV. Δυστυχώς ασκούνται και ισχυρές πιέσεις από παντού και σας όθησαν εσάς και τις υπηρεσίες σας να μην γίνουν σεβαστές ημερομηνίες. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα εφαρμόσετε αυτά που υποσχεθήκατε σύμφωνα με το Συμβούλιο Επιτήρησης που έλεγα πριν για να αποσυμφορηθεί κάπως η αγορά. Η ομάδα μας θα ήθελε οι προτάσεις σας να μας υποβληθούν ως έχουν και όχι με συνοδευόμενες από ερμηνείες. Επίσης, μας είπατε ότι θα κάνατε προτάσεις και για την επίλυση των κρίσεων. Τι έχει γίνει γι' αυτό, πότε θα ε, ε, δημοσιευθεί η πρότασή σας. Ναι, να επιβεβαιώσω, Σβεν Γιγκόλτ ότι είμαι θετικός και εργάζομαι επί μιας πρότασης για το θέμα των κινδύνων που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέτρα που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά προϊόντα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει δουλειά σε διεθνές επίπεδο για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να δούμε τις διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, και μαζί με τις υπηρεσίες μου κάνουμε μία αξιολόγηση, αλλά σας ε, επιβεβαιώνω τη δέσμευσή μου να παρουσιάσω ένα κείμενο για αυτό το ζήτημα. Και το είχατε ξαναναφέρει στην πρώτη μας συνάντηση, δεν το ξέχασα. Πιστεύω ότι εργαστήκαμε πολύ καλά με ικανές ομάδες επί του θέματος και προσπαθήσαμε να θέσουμε προτεραιότητες και ε, να θέσουμε προτεραιότητα στους ε, χρονικούς φορείς ε, γιατί μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι όπως ο τραπεζικός τομέας προκάλεσαν αυτή την κρίση. Εργάζομαι βέβαια και επί άλλων θεμάτων. Στον τομέα αυτό η προτεραιότητα είναι να θέσουμε σε εφαρμογή το solvency και το τελευταίο στάδιο θα είναι να εργαστούμε για τα θέματα που αναφερθήκατε για το θέμα της εξυγένσης. Για το σκιώδη τραπεζικό τομέα δεν θα περιμένετε πολύ, γιατί τον Ιούνιο θα παρουσιάσω την ανακοίνωση της Κομισιόν που θα συνοδευτεί και από νομοθετική πρόταση δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ για να εργαστούμε ε, και επί της πρότασης που αφορά τα market funds. Ε, βρισκόμαστε στο τελευταίο επίπεδο ε, ολοκληρωσής αυτής της πρότασης. Είναι έτοιμη και θα λάβει υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα ταμεία αλλά θα θέλαμε να καλύπτονται στην ε, περίπτωση του παράλληλου τραπεζικού τομέα. Θα θέλαμε και εκεί να διέπεται από διαφάνεια, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Επανέρχεται ο κύριος Γκίγκολτ. Δεν ήταν αυτή η ερώτησή μου. Η ερώτησή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Η SRB πρότεινε να απαγορευτεί η πρακτική του CNAV, Net Asset Value, πρακτικές ε, τέτοιες. Όμως η πρόταση ε, που έχει υποβληθεί δεν έχει ληφθεί υπόψη γιατί παρόλα που η CSRB πρώτη φορά πρότεινε να απαγορευτεί κάτι. Μπορείτε να μου βεβαιώσετε ότι εσείς θα υποστηρίξετε αυτή την πρόταση της ε, CSRB του Συμβουλίου. Επίτροπος, ε, εγώ ακούω πάντα τη γνώμη του Συμβουλίου πολύ προσεκτικά από τότε που ιδρύθηκε. Ξέρω την ανησυχία σας και θέλετε να απαγορευτούν κάποιες δραστηριότητες, να καταπολεμηθούν. Εγώ λαμβάνω υπόψη τις απόψεις του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και ε, μπορώ να σας πω ότι το κείμενο είναι σχεδόν έτοιμο. Απλώς ε, σας ζητώ να σεβαστείτε την άποψη του που εκφράζω. Και εγώ πρέπει να σεβαστώ τη δουλειά όλου του Σώματος των Επιτρόπων. Δεν μπορώ να σας πω κάποια πράγματα δημόσια εδώ σήμερα, δηλαδή για αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε συζητήσει ακόμη. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου έχει σχέση με το θέμα των καταθέσεων και με την προτινόμενη οδηγία για την ανακάψη και την εξυγίαση των τραπεζών. Θα χρησιμοποιήσω το ερώτημα που ακούγεται στην Ελλάδα, που ακούγεται στην Ελλάδα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πριν από την κρίση ήταν από τα πιο ασφαλή και τα πιο υγιή διότι δεν ήταν εκτεθειμένο σε τοξικά επενδυτικά προϊόντα και επίσης τα δάνεια που έδιναν είχαν καλή ποιότητα εγγύησει Μετά από το κούρεμα των κρατικών ομολόγων, μετά από την αύξηση της εξόδου των κεφαλαίων ε, ε εκτός Ελλάδας και την πτώση των αξιών αποφασίστηκε να δοθεί το ποσό των 50 δις για την ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Ε, αυτά όμως τα μεγέθη κύριε Επίτροπε ήταν με τα δεδομένα των αρχών του 2012. Έκτοτε όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά υπάρχει μια εντυνόμενη ύφεση στην Ελλάδα με συνεπακόλουθο, με αποτέλεσμα δηλαδή, να αυξάνεται ο όγκος και ο αριθμός των επισφαλών δανείων, των κόκκινων δανείων και επομένως υπάρχει μια πρόσθετη ανησυχία. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν το έχετε υπόψη σας και αν έχετε κάτι παραπάνω να μου πείτε όσο αφορά αυτό τον κίνδυνο που προσθέτει ανησυχία όσο αφορά το τραπεζικό σύστημα ε, και βεβαίως στην περίπτωση που ξεφύγει αυτή η κατάσταση με συνεχιζόμενο τον όγκο της Μάζα, των κόκκινων δανείων τι μπορεί να γίνει, ποιος μηχανισμός θα κινητοποιηθεί, θα εφαρμοστεί η οδηγία από τώρα σε σχέση με το κούρεμα των καταθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χουντή μου, κατανοώ τι εννοείται και τις ανησυχίες σας που είναι παρόμοιες με των Ελλήνων επιχειρηματιών και των πολιτών στους οποίους ζητάνε όλο και περισσότερες προσπάθειες. Εγώ ως Επίτροπος υπεύθυνος για τη ρύθμιση του δημοσιονομικού και χρηματοπιστικού τομέα δεν ξέρω τι να σας απαντήσω γιατί τα κείμενα που ετοιμάζουμε απαιτούν το καθένα πολύ καιρό, πάνω από χρόνο για να εγκριθούν και να εφαρμοστούν. Δεν πρόκειται λοιπόν να διορθώσουν τα κακό κείμενα του παρελθόντος ή τις ζημίες του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να αναστρέψουμε το χρόνο και να λύσουμε προβλήματα δημοσίου ελλείμματος του παρελθόντος ή την τοξική σύνδεση μεταξύ κρατικού χρέους και τραπεζικής κρίσης, την έλλειψη, της έλλειψης εποπτείας κλπ. Αυτά τα κείμενα θα χρησιμοποιηθούν για μερικούς από τώρα, όχι πολλούς, πολλά, όχι πολλά μάλλον, και τα περισσότερα από αύριο και εσείς το εξετάζετε βέβαια και με βάση τα μαθήματα της προηγούμενης φάσης της κρίσης προσπαθούμε να διορθώσουμε το μέλλον, όχι το παρελθόν. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα, θα μπορούσα να μιλήσω και για την κρίση στην Κύπρο ή στην Ιρλανδία ή στην Ισπανία, τα εξετάζουμε ένα-ένα είτε πρόκειται για την επιτήρηση εποπτεία, είτε για τη διακυβέρνηση, είτε για την ανακεφαλαιοποίηση. Όλα αυτά τα νομοθετήματα βασίζονται στα μαθήματα από το παρελθόν. Αν είχαν εφαρμοστεί τέτοιοι νόμοι προηγουμένως, οι περισσότερες τραπεζικές κρίσεις που ζήσαμε με την πλάτη στον τοίχο εδώ και 4-5 χρόνια θα τις είχαμε αποφύγει ή ελέγξει πολύ καλύτερα. Θα αναφέρω στον συνάδελφό μου όλοι ρεν τις ανησυχίες σας. Ίσως να μπορούσα να πω ότι στις προσπάθειες που ζητούμε από πολλές χώρες για σταθεροποίηση δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική και τραπεζική, εγώ προσωπικά ως επίτροπος εδώ και αρκετό καιρό τονίζω την ιδέα της διαφοροποίησης ενός κατάλληλου ρυθμού για τις προσπάθειες ώστε η λιτότητα σε ορισμένες χώρες να μην καταλήξει σε μηδενική ανάπτυξη. Τα έσοδα δηλαδή να μην μειώνονται περισσότερο από ότι οι μειώσεις των εξόδων λειτουργίας. Γι' αυτό ζητώ πάντοτε διαφοροποιημένη αντιμετώπιση και προσαρμογή στο ρυθμό της κάθε χώρας που απαιτείται στην κάθε χώρα. Ο Παύλος. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, είπατε ότι η εποπτεία οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ μαζί σας, όμως για να συνεχίσει να ισχύει κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν ο δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης. Είπατε ότι τον Ιούνιο θα παρουσιάσετε μία ενιαία πρόταση για το Ταμείο της Εξυγίανσης των Τραπεζών. Χαίρομαι που ακούω αυτή την είδηση, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε θετικό μήνυμα στις αγορές, αλλά και στους πολίτες, ότι οι πολιτικοί εργαζόμαστε για την έξοδο από την κρίση για να μην επαναληφθεί αυτή η κρίση. Παρ' όλα αυτά, κάποια κράτη-μέλη έχουν δείξει δισταγμού απέναντι στην αναγκαιότητα ή μη να αλλάχθουν οι συνθήκε για να εφαρμοστεί ο δεύτερο πυλώνας τη Τραπεζική Ένωση. Δεδομένη τη σημασία των καιρών, πιστεύετε ότι θα είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι συνθήκες ε, για να εφαρμοστεί ο δεύτερο πυλώνας τη τραπεζική Ένωση. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρνιά. Η απάντηση μου είναι όχι. Πιστεύω ότι μπορούμε και πρόκειται να παρουσιάσουμε την πρόταση ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εξυγίανσης βασιζόμενη στις σημερινές συνθήκες. Και εγώ επ' αυτής της βάσης εργάζομαι, αποκοινούμε τους συναδέλφους και φυσικά με την υποστήριξη και των νομικών μας υπηρεσιών. Και φυσικά σε συνεργασία και με το Συμβούλιο και με τις υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Κύριε Σάλμπα, κατανοώ τις ανησυχίες που εκφράζονται από κάποιες χώρες, ιδίως από τη Γερμανία. Πάντοτε ακούω, ιδίως όσα λέει ο κ. Σόιμπλε, με πολύ προσοχή και σεβασμό. Η Γερμανία έχει μία ανησυχία που την κατανοώ και δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Είναι της ασφάλειας δικαίου των όσων κάνουμε. Και έχει και δικές της ανησυχίες που σχετίζονται με το δικαστήριο της Καλζούης και για το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός του χρόνου. Γι' αυτό δεν απορρίπτω την ιδέα. Αφού θα έχει τεθεί σε λειτουργία το σύνολο της Τραπεζικής Ένωσης, η υποπτία, ο μηχανισμός εξυγίανσης, όπως είναι δυνατόν να γίνει στο πλαίσιο της σημερινής συνθήκης, μια στοχευμένη τροποποίηση της συνθήκης, σε μετέπειτα στάδιο θα μας επέτρεπε να παγιώσουμε ακόμη καλύτερο το σύστημα. Όμως εγώ κατανοώ την ανησυχία της Γερμανίας και την κατανοώ ε, ακόμη καλύτερα όταν η Κομισιόν ε, στο blueprint, ε, στο μοντέλο πρότεινε ότι για να λειτουργήσει καλύτερα η Οικονομική και Μεσοματική Ένωση πρέπει να υπάρχει τροποποίηση τη συνθήκη. Εμεί οι ίδιοι, δηλαδή η Κομισιόν προτείναμε τροποποίηση συνθήκη. Δεν πούμε λοιπόν σήμερα ότι δεν είναι κάτι τέτοιο χρήσιμο ή δυνατό, όμως είναι δυνατό να λειτουργήσει το σύστημα στο σημερινό καθεστώς και θα μπορέσουμε να ε, το βελτιώσουμε και να το παγιώσουμε με μια μετέπειτα τροποποίηση της συνθήκες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Θα ήθελα να πω ότι αρκετές ερωτήσεις που ήθελα να κάνω ετέθησαν ε, και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα θέμα πρόκειται για το τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ΦΕΔ, κύριε Επίτροπε, δημοσίευσε στοιχεία με βάση τα οποία οι αλλοδαπές ε, τράπεζες ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι μεδαπές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό όμως ε, σημαίνει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αλλοδαπών τραπεζών και κυρίως και η δαιμονία των αλλοδαπών τραπεζών στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εσείς ως αρμόδιος επίτροπος ταχτήκατε κατά αυτού του πρόδειλου προστατευτισμού. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει τι θα γίνει τελικά, πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 και πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σημαντική ερώτηση όπως συνήθως από τον συνάδελφο αυτό. Αφορά την ε, αξιοπιστία του τι θα αποφασίσουμε μαζί στο Z20. Υπενθυμίζω ότι είχαμε αποφασίσει ήδη για την ε, ευστάθεια του τραπεζικού τομέα να εφαρμόσουμε τις περισσότερες από τις συστάσεις του z 20 Ο Ομπάμα, ε, όλοι οι άλλοι ήταν παρόντες. Και εγώ δίνω μεγάλη σημασία στην αξιοπιστία του Z20 για τις πιο αποτελεσματικές διεθνείς δοσοληψίες. Όχι πάντοτε με τους ίδιους κανόνες και νόμους, αλλά παράλληλα να εφαρμόζουμε ανάλογη νομοθεσία για ανάλογους τομείς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τραπεζικό τομέα. Γνωρίζω καλά το πρόβλημα που αναφέρατε που με έχει οθήσει εξάλλου να απευθυνθώ στις Αμερικανικές Αρχές και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του ΦΕΔ και στην τελευταία μου επίσκεψη στις ΗΠΑ είχα μια χρήσιμη συνάντηση και με τον κύριο Τάουλο και με τον Τζακ Λό, τον νέο υφυπουργό, υπουργό οικονομικών και άλλοι Ευρωπαίοι Υπουργοί αλλά και ο Καναδός, ο Ιάπων Υπουργοί Οικονομικών με στήριξαν τις απόψεις μου γιατί είπα ότι τα μονόπλευρα μέτρα που θέλουν να εφαρμόσουν οι Αμερικανοί στις ξένες τράπεζες που λειτουργούν στη ΣΥΠΑ μέσω του νόμου σχεδίου που λέγεται Foreign Banking Organizations για μας είναι όχι μόνο μονόπλευρα αλλά και άνηση μεταχείριση και θα βλάψουν και τις ξένες αυτές τράπεζες και τις αμερικανικές. Γιατί δεν πρέπει να αυταπατώμαστε, να λέμε την αλήθεια. Αν υπάρξουν μέτρα άνησης μεταχείρισης θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και τα λέω αυτά γνωρίζοντας τι λέω. Δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα. Γιατί πρέπει να βρούμε μεθόδους και μέτρα ισότιμα την 8 μου επίσκεψη στις ΗΠΑ τον Ιούλιο θα την κάνω για να δούμε ακριβώς ποιες μπορεί να, ποια μέτρα μπορεί να έχουν ισότιμες εξισωμένες επιπτώσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης με επικοδομητικό λοιπόν πνεύμα αλλά χωρίς αφέλεια θα κάνω αυτές τις συναντήσεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε υπερβάνς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Γι' αυτό το τελευταίο. Έχω μεγάλες ανησυχίες για αυτήν τη διάσταση της συμφωνίας είπα ένωσης, όχι για την εμιβαιότητα. Αυτό φαντάζομαι όλοι το ξέρουν και τη συμφωνούν, αλλά η συμφωνία αφορά και τις επενδύσεις, μια μεγάλη αγορά επενδύσεων, ενώ πολλές αμερικανικές επενδύσεις, τις λέμε επενδύσεις αλλά θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε και αλλιώς, είναι σε θέση να κάνουν όμοιρο την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Όταν ο Goldman Sachs γονατίζει την Ελλάδα, γιατί να πούμε ότι με τέτοια μέτρα θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το στρατηγικό αυτό πρόβλημα. Οι Αμερικανοί επενδυτές μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να κάνουν τέτοια πράγματα. Σας προτείνω ακόμη μία από τις συστάσεις που περιοδικά σας κάνω ότι η ICC είναι πιο ανεξάρτητο όργανο από την ΕΚΤ. E για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας, όλοι νομίζω ή πολλοί τουλάχιστον ανέμεναν με ανυπομονησία το έγγραφό σας. Δεν ξέρω αν είναι διαθήκη ή κληρονομιά, θα θέλαμε όμως το έγγραφο αυτό να είχε γραφτεί στην αρχή της διαδικασίας, όχι στο τέλος, γιατί όταν δούμε, αν δούμε τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση. Τελικά πρέπει τον κατάλογο που γράψατε από χρόνο σε χρόνο, τη Βασιλεία 2 ή τα υπόλοιπα, να τα ξαναδούμε πρέπει από την αρχή. Αλλά δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί η ιστορία ή θα γραφτεί α, αλλιώς και άλλη φορά. Όχι, μια στιγμή, την ερώτησή μου τελειώνω. Εγώ είμαι η μόνη που την κόβεται. Μα είστε οι μόνοι που ξεπερνάτε τα δύο λεπτά γι' αυτό. Εγώ είπα δύο λεπτά. Λίγο, λίγο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μου ερώτημα είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε τα πράγματα, να συνδέσετε αυτά που κάνει ο συνάδελφός σας σε μέτα με αυτά που θέλετε εσείς. Αν θέλετε να επιδείξετε συνέπεια και εσείς και εμείς, η χρηματοδότηση της οικονομίας ή των μακροπρόθεσμων επενδύσεων προϋποθέτει ότι στη φορολόγηση της, της αποταμίευσης θα συνδυαστούν οι μεσοπρόθεσμοι με τους μακροπρόθεσμους στόχους και αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πολίτες. Μάλιστα. Η κυρία Μπερέση καταρχήν αναφέρθηκε στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Ήμουν στον Άσικτον την επόμενη μέρα της ομιλίας του Πρόεδρου Ομπάμα για όπου αναφέρθηκε σε αυτή την συμφωνία και είπε ότι θέλουμε αυτή την παγκοσμιτερική σχέση fair and free, δίκαιη και ελεύθερη. Αυτές ήταν οι δύο λέξεις του Πρόεδρου Ομπάμα και έτσι λοιπόν να μην λέμε ότι είναι μόνο ελεύθερη αλλά και δίκαιη, το είπε και ο Πρόεδρος Ομπάμα και ε, ο συνάδελφος συζητά τώρα το θέμα με το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στη συμφωνία είτε μιλάμε για τη διεύρυνση της πρόσβασης είτε για το κανονιστικό πλαίσιο. Στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν θεσμικοί λόγοι βέβαια που ε, καθορίζουν ε, ε, το ρόλο των αρμοδίων αρχών. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργό Εμπορίου Παραδείγματο Χάρη δεν μπορεί να μιλήσει εξ ονόματό του, όμω εμεί θέλουμε να έχουμε μία αυστηρή στάση στις διαπραγματεύσεις και να δημιουργήσουμε ίσους κανόνες για όλους και να έχουμε και ρυθμίσεις για την πρόσβαση. Καθώς με αναφερθήκατε στην Goldman Sachs και σε άλλα προβλήματα, να υπενθυμίσω ότι έχουμε εργαλεία, καινούργια εργαλεία για να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά τα κείμενα που θα ενισχύσουμε και με τη δική σας συνεισφορά για την καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών, ε, για τις καταχρήσεις ε, των αγορών, ε, ποινικοποιούμε μάλιστα και ορισμένες πρακτικές και έχουμε και το νέο στοιχείο την ύπαρξη της εποπτικής αρχής που θα υπάρχει στην Ευρωζώνη. Αυτό θα αλλάξει πάρα πολλά. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία και για τις, τα αλλοδαπά υποκαταστήματα, τις αλλοδαπές έτσι, λοιπόν, εγώ εδώ, αν μου επιτρέπετε, ε, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα για το μέλλον ε, και τώρα εδώ δεν υπογράφω διαθήκη, αλλά εδώ ε, να σας πω ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2010 είπα ότι έπρεπε να δούμε τα διδάγματα της κρίσης και είχα μπροστά μου όλη την ατζέντα της G20 και ε, εγώ μαζί με τις ομάδες μου δεν σας ε, κάλεσα απλώς να κάνουμε μια συζήτηση αφηρημένη, αλλά σας ανέφερα πώς ε, θα εφαρμοστούν οι κανόνες της G20 σε όλους τους τομείς, σε όλες τις αγορές και σε όλα τα προϊόντα. Σταματώ εδώ. Επειδή θα φύγει ο Επίτροπος, στις 6 και 4 έχουμε τώρα δυσκολίες με το χρόνο. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει τώρα να περιορίσω τις ερωτήσεις στο ένα λεπτό και να έχουμε απαντήσει στα δύο λεπτά. Και Περβάνς δεν μπορείς ε, να καταχράσει το χρόνο που σου δίνουμε σε αυτή την επιτροπή. Εσύ εδώ καταχράσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φέιου. Σας ε, συγχαίρω για όλο το έργο σας και πολύ γρήγορα να θέσω δύο ερωτήσεις. Έχουν να κάνουν με το τραπεζικό ζήτημα. Μετά το πρόβλημα που είχαμε στην Κύπρο, αισθανθήκαμε μία έλλειψη εμπιστοσύνη από τους πολίτες ε, στο τραπεζικό σύστημα και φυσικά αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη εμπιστοσύνη των καταθετών. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε τι εγγυήσει ε, θα δώσετε στους ε, πολίτες ε, που έχουν τις καταθέσεις τους σε κράτη που μπορεί να αισθανθούν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με λύσεις που θα μας οδηγήσουν στο να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τη διάσωση των τραπεζών αναφερθήκατε στην εγγύηση καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω με τις επιχειρήσεις ε, που πολλές φορές ε, έχουν έλλειψη λευστότητα για να πληρώσουν ε, τους μισθούς το χάρη. Τι θα γίνεται. Λέω στον κύριο Φέιο ότι σε καμία στιγμή στο μυαλό μου ο τρόπος που δράσαμε σε κατεπίγουσες συνθήκες ε, με την ε, νέα Κυπριακή Αρχή ε, πριν ξεσπάσει η Κυπριακή κρίση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μοντέλο για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ανανομοθέτημα με την Τραπεζική Ένωση στην Ευρωζώνη είναι για τις 27-28 χώρες της Ευρώπης ε, να ε, υπάρχει ε, ένα σύστημα σαφές με την Τραπεζική Ένωση και το σύστημα τραπεζικών εγγύσεων. Ένα σύστημα λοιπόν που θα είναι διαφανές και θα έχει ανακοινωθεί από την αρχή. Δεν ίσχυε κάτι τέτοιο στην Κύπρο, ενώ τώρα όλοι θα ξέρουν τι θα περιμένουν αν η τράπεζα στην οποία κάποιος είναι μέτοχος πιστωτής καταθέτης βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως η Κύπρος ε, δεν αποτελεί μοντέλο, Πρόκειται για ε, τη διαχείριση πολύ, μιας πολύ δύσκολης κατάστασης ε, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Όμως σε ό,τι αφορά τους καταθέτες, να σας πω ότι κάτω από τις 100.000 θα υπάρχει απόλυτη προστασία για τις καταθέσεις άνω των 100.000. Εγώ ο ίδιος Ζήτησα και τώρα, συζητάμε το θέμα του συμβιβασμού στον τραμερή διάλογο, να υπάρχει μία προτίμηση για ε, τους καταθέτες ε, πάνω από τους 100.000 που θα κληθούν τελευταίοι στον κατάλογο. Και επίσης ε, έχουν ζητηθεί κάποιες εξαιρέσεις για τα νοσοκομεία, για φιλανθρωπικά ιδρύματα, θα ήθελα αυτός ο κατάλογος των εξαιρέσεων των όσων καλούνται να καλύψουν ένα μέρος ε, του κόστους ε, της κατάρρευσης τράπεζας να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένων. Θέλουμε να προστατεύσουμε φυσικά τις μικρές και ζωές επιχειρήσεις και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, αλλά θέλουμε να είναι πολύ πλαισιωμένη αυτή η λίστα και πολύ περιορισμένη. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα ήρθατε εδώ για να μας απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Ε, καταλαβαίνετε ότι εγώ θα ήθελα μια ε, καλύτερη απάντηση από αυτή που μου δώσετε προηγουμένως για την εξασφάλιση των καταθέσεων. Ξεκινήσαμε με την Τραπεζική Ένωση και καταφέραμε δύο πολύ καλά πράγματα, αλλά διαπιστώνω ότι και εσείς ε, στη σημερινή συζήτηση περιορίζετε για δύο μόνο πράγματα όσον αφορά τις τράπεζες. Μιλάτε για την αναδιάρθρωση, για το Ταμείο Εξυγένσης ε, και ε, την, ε, και άλλα παρεμφερή θέματα, όμως όχι για την εξασφάλιση των καταθέσεων. Εγώ όμως πιστεύω ότι αν δεν μπορέσουμε να νομοθετήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών που τη χάσαμε μετά το χάος ε, της ε, Κύπρου. Στη Γερμανία οι σπιουμετρήσεις λένε το 70% των καταθέσεων πίστευαν ότι οι καταθέσεις τους δεν είναι ασφαλείς και μετά... Ε, 14 ημέρες μετά την Κύπρο μόνο το 34% πίστευαν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή στις γερμανικές τράπεζες. Εγώ πιστεύω μόνο αν ολοκληρώσουμε την ε, νομοθεσία περί καταθέσεων θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών. Η Κομισιόν πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά σε αυτή την τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Κοιτάξτε, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας για το κείμενο για τις εγγυήσεις των καταθέσεων που για είναι τμήμα του μηχανισμού σταθεροποίησης του τραπεζικού τομέα και που συζητιέται με βάση την πρότασή μου εδώ και περίπου δύο χρόνια για να καταλήξει τελικά εκεί που ξέρετε. Δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε για την Κύπρο πολύ ώρα, αλλά εκείνο το Σαββατοκύριακο που δόθηκε η εντύπωση ότι θα φορολογούσαμε τις μικροκαταθέσεις αυτό ήταν παρεξήγηση και δείχνει ακριβώς ότι υπήρχε έλλειψη εμπιστοσύνης γιατί υπήρχε η οδηγία για την εγγύηση των μικροκαταθέσεων και φάνηκε σαν να μην τη σεβόμαστε. Η Συμφωνία λοιπόν αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Τραπεζών σέβεται την οδηγία εκείνη και συμφωνώ ότι τώρα πρέπει για να ξαεπανέλθουμε στην εμπιστοσύνη να αναδομηθεί το όλο σύστημα που βασίζεται στα δύο κείμενα εγγύηση των καταθέσεων και το ψήφισμα του Γκούναρ Χόκμαρκ και για την Ευρωζώνη την Τραπεζική Ένωση που θα συνδυάζει την εποπτεία που έχει ήδη ετοιμαστεί και το ψήφισμα για το οποίο θα συζητήσουμε προκαταρκτικά την επόμενη εβδομάδα μέχρι να καταθέσουμε μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Συμφωνώ όμως ότι χρειάζονται όλα αυτά για να επανέλθει η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε. Βέρνος Λέων. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πολλή δουλειά σας. Ο δρόμος ε, για την σταθεροποίηση ευρωζώνης και τις ε, ρυθμίσεις είναι ακόμα μακρύς. Καταρχήν, ε, όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό ΕΜΙΡ, κυρίως όσον αφορά τις μη χρηματοπιστωτικές εξασφαλίσεις από παράγωγα. Δεύτερον, ε, τελικά, τι θα γίνει με την πρότασή σας για τη ρύθμιση των σκιωδών τραπεζών, πότε πρόκειται να την καταθέσετε και τρίτον, ε, τι ακριβώς, ε, πώς μπορεί να συμβιβαστεί ο, ο μηχανισμός εξυγίανσης με, τις, με τον ανταγωνισμό. Τέλος, όσον αφορά την σύνταξη γύρατος, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν προτίθεστε να επιβάλλετε περαιτέρω όρους στα συνταξιωτικά ταμεία, γιατί κυριότερο στόχος σας είναι να τα σταθεροποιήσετε. Συγγνώμη, Βέρνερ, αλλά δεν κατάλαβα το τελευταίο τμήμα της ερώτησης. Κοιτάξτε, να το εξηγήσω λιγάκι. Αναφέρομαι στα συνταξιωτικά ταμεία και στα επικουρικά ταμεία. Ε, τι θα κάνετε, θα εκπονήσετε μόνο διατάξεις διαφάνειας ή προτίθεστε να καταστήσετε τις υπάρχουσες διατάξεις ακόμα πιο αυστηρές. Για το θέμα των διεθνών διαπραγματεύσεων που σχετίζεται με τον κανονισμό ΕΜΗΡ να απαντήσω και σε μια προηγούμενη ερώτηση για το που βρισκόμαστε και για το τι πρέπει να γίνει κάποια δουλειά όχι μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών μόνο αλλά και στο πλαίσιο της ομάδας των αριθμιστικών αρχών που θα συνεδριάσει στις 29 Μαΐου στο Χανκόνγκ. Είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις αυτές ακριβώς λόγω της θέσης της EFTC και στις αρχές ε, ε, Ιουλίου θα συναντηθώ με τον πρόεδρο της FTC για αυτό το θέμα, για το shadow banking. Θα υλοποιηθεί η πρόταση και θα συνοδεύεται με μία πρώτη νομοθετική πρόταση, όπως είπα, τον Ιούνιο. Θα έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση και την πρώτη νομοθετική πρόταση. Επιβεβαιώνω ότι για τα συντοξιδετικά ταμεία και για τα ε, επαγγελματικά επικορικά ταμεία που είναι μεταξύ των κύριων φορέων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της οικονομίας. Έχουμε προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα που αφορούν την υποδομή, τα δίκτυα, την εξάρτηση, την οικολογική μετάβαση. Θα είμαι πολύ προσεκτικός στις επιλογές που θα κάνω για να παρουσιάσω πριν από τα τέλη του έτους ε, μία πρόταση νομοθετήματος ε, για τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την εποπτεία των συνταξιδοτικών ταμείων και να αφήσω για αργότερα το θέμα των κανόνων προληπτικής εποπτείας και αφαιρεγγιότητας γιατί δεν έχω τα χρήσιμα συγκεκριμένα και αντικειμενικά στοιχεία για να αποφασίσω ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας, Μέδερετ Φρακφούρτη, μου είπε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να κάνει αυτή την αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν, επειδή εγώ δεν παίρνω αυθόρμητες αποφάσεις, προσπάθησα να διακρίνω αυτά τα δύο μέρη και κατά τη διάρκεια της ιτίας αυτής της Κομισιόν να δώσω προτεραιότητα στο θέμα της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της εποπτείας των συνδεξιδοτικών ταμείων και να δούμε αργότερα το θέμα των εποπτικών μέτρων και της φερεγγιότητας. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Κοιτάξτε, μπορούμε να ρωτήσουμε αύριο, αν θέλετε, τον Επίτροπο κύριο Αλμούνια. Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο. Στην περίπτωση Τέξια Μπάνκια και Μπέ, ε, την αναδιάρθρωση την έκανε ο Επίτροπος Αρμόδιο για τον Ανταγωνισμό. Εσείς τι πιστεύετε, στο μέλλον θα διατηρήσει τις θέση του αυτός Επίτροπος ή θα τις χάσει. Η απάντηση μου είναι ναι. Πόση επιτυχία θα είχα αν ναι, μετά από όλε αυτέ τι μεταρρυθμίσει έλεγα δεν υπάρχει πλέον δουλειά για τον επίτροπο ανταγωνισμού. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Όχι, όχι, θα υπάρχουν ακόμη κρατικέ πολιτικέ και θα υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου θα χρειαζόμαστε χρηματοδότηση από το δημόσια κονδύλι. Έτσι λοιπόν οι κρατικοί κανόνες θα συνεχίσουν να ισχύουν και ο Επίτροπος ε, αρμοδίζει τον ανταγωνισμό θα έχει ακόμη πολλή δουλειά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ε, δεν μπορούμε να γνώσουμε τις συνθήκες με τις ε, οδηγίες που εκπονούμε. Τις τρεις τελευταίες ερωτήσεις θα τις πάρω από κοινού Άννη Όλοι Σμιτ, ένα λεπτό παρακαλώ ο καθένας. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, σας παρακαλώ πολύ. Ε, μην μιλάτε και δώστε μια ευκαιρία στους ε, συναδέλφους ε, να μιλήσουν. Η Άννη λοιπόν, μετά όλοι και μετά ο Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπο. καλημέρα. Φαντάζομαι παρακολουθείτε τις δύσκολες συζητήσεις στο Συμβούλιο Μεταξύ των 11 χωρών που αποφάσισαν να συνεχίσουν στην εφαρμογή της ενισχυμένης με την ενισχυμένη συνεργασία στην εφαρμογή του νόμου των δοσοληψιών των συναλλαγών. Διαπιστώνουμε και προσπάθειες των επιχειρήσεων της βιομηχανίας να δαιμονοποιήσουν τον φόρο αυτόν και να αποδυναμώσουν την πρόταση. Ερωτώ λοιπόν, συμμερίζεστε ή όχι τις ανησυχίες που έχουν ακουστεί, είστε παραμένετε υπέρ του φόρου αυτού ή είστε από εκείνους που λένε ότι ο φόρος ίσως να έχει να... να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στην δημοσιονομική χρηματοπιστωτική δραστηριότητα. Ή αντίθετα θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλλει ο φόρος αυτός σε μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Κυρία Ποτηματά. Α, όχι, όχι, περιμένετε να απαντήσετε και τις τρεις ερωτήσεις. Έτσι είναι πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Η Ρώδη Κράτσα. Μα πολλές μαζί γιατί δεν θα προλάβει αλλιώς ο Επίτροπος. Κύριε Επίτροπε, ε, παίρνω ευκαιρία από αυτό που είπατε ότι οι ανησυχίες για το τραπεζικό σύστημα δεν είναι θεωρητικές και από αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου για τι τις ανησυχίες που εξέφρασαν για το θέμα των καταθέσεων και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη πτυχή σύντομα. Ε, υπάρχει περίπτωση η ανασφάλεια να αυξηθεί στις χώρες της περιφέρειας με τα περισσότερα προβλήματα και να υπάρχει μετακίνηση ε, κεφαλαίων προς τις τράπεζες του κέντρου και με τον τρόπο αυτό να αυξηθούν και οι ανισορροπίες και τα προβλήματα στην περιφέρεια μέσα στη διαδικασία του bail in. Ε, υπάρχει κάποιος μηχανισμός, κάποιο σχέδιο που αντιμετωπίζει αυτή την ανασφάλεια και την ανισορροπία που μπορεί να δημιουργηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Thank ε, κύριε Επίτροπε, εσείς ε, υποσχεθήκατε όταν πρωτοήρθατε εδώ να επιβάλλετε ρυθμίσεις και το κάνατε αυτό, καμία εμφιβολία. Όμως ε, πριν φύγετε από το αξίωμά σας, μήπως μπορείτε να υποσχεθείτε ότι θα έχετε και ένα συνολικό, μια συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων. Εμείς ε, είμαστε υπόλογοι ε, απέναντι στους πολίτες και στις ε, χρηματοψηφιακές αγορές. Μπορείτε λοιπόν να υποσχεθείτε ότι πριν ολοκληρωθεί η θητεία σας θα ρυθμίσετε αυτά τα οποία είχατε υποσχεθεί ο κύριος Επίτροπος τρεις ερωτήσεις και τρεις τηλεγραφικές απαιτήσει. Αλλά φυσικά, Πρόεδρε, μπορώ να επανέλθω για να συνεχίσουμε το διάλογο. Κυρία Αποδηματά, μου έθεσε το θέμα του φόρου χρηματοπιστωτικών συνέλεγων. Δεν έχω αλλάξει θέση. Πιστεύω ότι αυτό το φόρο, έτσι όπως προτάθηκε από την Κομισιόν, όπως συμμετέχω, είναι τεχνικά εύκολος να εφαρμοστεί, οικονομικά βιώσιμος και πολιτικά δίκαιος. Είναι δυνατό στο περιθώριο να διορθωθεί η βάση αυτού του φόρου, όμως τώρα στο Συμβούλιο των Υπουργών είναι αυτό που θα πάρει τις ευθύνες, που θα αναλάβει τις ευθύνες του, όμως τεχνικά είναι εύκολο να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος ε, και μπορεί να είναι βιώσιμος οικονομικά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά για τις χρηματαγορές, οι φορολογούμενοι έχουν πληρώσει πολύ για τις χρηματαγορές, επομένως είναι βιώσιμος και είναι και ηθικά και πολιτικά δίκαιος κυρία Κράτσα, να υπάρχει ένας κίνδυνος κατακαιρματισμού εντός της ενίας αγορά. Είμαι πολύ προσεκτικό για το θέμα αυτό, γιατί πέρα από τα συγκυριακά μέτρα που θα μπορούσαν να, να ληφθούν και που ελήφθησαν μάλιστα σε κάποιες χώρες από κάποιες αριθμιστικέ αρχές, διασφαλίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων εντό τη ενίας αγορά. Και αυτό που κάνουμε με όλα τα μέσα ε, που εκπονήσαμε ακριβώς ήταν να περιορίσουμε τον κίνδυνο του κατακαιρματισμού στον οποίο αναφερθήκατε. Όμως ε, δεν έχει περάσει εδώ και πολύ καιρό που το διατραπεζικό σύστημα ήταν εντελώς μπλοκαρι, μπλοκαρισμένο. Ε, υπήρξε ουσιαστικά επανεθνικοποίηση των ε, κυκλωμάτων ρευστότητα και χάρη σε μία ριζική απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, θέσαμε σε νέα κίνηση το διατραπεζικό σύστημα. Έτσι λοιπόν εγώ νομίζω ότι μπορούμε να περιορίσουμε αυτόν τον κίνδυνο κατακαιρματισμού και να πω στον κύριο Σμιτ ότι η απάντησή μου είναι ναι. Ναι. Μου φαίνεται λογικό Τώρα που πάνω κάτω γνωρίζουμε την αρχιτεκτονική αλλά και το περιεχόμενο των νόμων αυτό, που διαφέρει από αυτό που είχαμε φανταστεί στην αρχή, όταν κάποια κείμενα βρίσκονταν απλώς στη λίστα της G20, παραδείγματος χάρη Βασιλεία 3. Έτσι λοιπόν μου φαίνεται τώρα να πολύ λογικό να ανακοινώσω ότι θα έχουμε μια τέτοια καθολική μελέτη αντικτύπου, γιατί δεν είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Και πριν τρία χρόνια σας είχα πει ότι πρέπει να υπάρχουν υγιείς βάσεις για τις χρηματαγορές. Και φυσικά κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αγορές και σε αυτό το πνεύμα εργάζομαι εγώ. Ωραία, πρέπει να φύγει στο Άμστερνταμ ο Επίτροπος. Αύριο στις 10 αρχίζουμε.